Καλημέρα σε όλους μας. Ας αρχίσουμε. Σας θυμίζω ότι το Σάββατο πέθανε ο διευθυντής ε, της Όλαφ, ο κύριος Μπρούνερ και εξ ονόματός μου ως πρόεδρος της Επιτροπής Ελέγχου του και εκ μέρους όλων των μελών θεωρώ και εκ μέρους των άλλων δύο επιτροπών που σήμερα παρίστανται εκφράζουμε τα θερμά μας συλληπιτήρια στην οικογένεια του κυρίου Μπρούνερ μέχρι το τέλος δούλεψε προσπαθώντας να φέρει σε πέρας με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το έργο του στην Όλαφ. Καλωσορίζω τον υποψήφιο επίτροπο, κύριο Σεμέτα. Θα είναι μαζί μας τρεις ώρες σήμερα στη σημαντική ακρόαση. Τον ευχαριστώ. Επίσης καλωσορίζω και τους άλλους συναδέλφους, τους πρέδους της ΣΥΜΚΟ και της ΕΚΟΝ, του κύριο Άρμπουρ και τη Συρία Σεραμπόλσκα. Επίσης ε, καλωσορίζω και τους συναδέλφους της Επιτροπής Ελέγχου Προπολογισμού και των άλλων δύο επιτροπών. Με βάση τον κανονισμό θα κρίνουμε τον Επίτροπο με βάση τις γενικές δεξιότητες του, την δέσμευσή του και την ε, ανεξαρτησία από διαφόρων ειδών υποχρεώσεις. Όπως ξέρετε, ο Επίτροπος ήδη απάντησε γραπτά στις πέντε ε, ερωτήσεις που τετέθησαν στο ερωτηματολόγιο. Οι απαντήσεις υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες. Επίσης, το βιογραφικό σημείωμα, η δήλωση των οικονομικών συμφερόντων, το mission statement του κ. Σεμέτα και την επιστολή του Πρόεδρου Μπαρόσο, μόνο στα αγγλικά. Πρέπει να τηρήσουμε το χρονοδιάγραμμα σήμερα. Ο υποψήφιος επίτροπος, μετά την εισαγωγή μου, θα έχει 10 λεπτά χρόνο μετά 2 ώρες και 45 λεπτά ερωτήσεις με βάση τις πολιτικές ομάδες. Πρέπει απολύτως να σέβεστε το χρόνο, διαφορετικά θα σας διακόπτω ένα λεπτό η κάθε ερώτηση, δύο λεπτά η απάντηση του Επιτρόπου και μία, ένα λεπτό η δευτερολογία, αν θέλει ο βουλευτής, και ένα λεπτό η δευτερολογία του υποψηφίου. Τέλος, υπάρχει δυνατότητα μια σύντομη δήλωση 10 λεπτών εκ μέρους του ε, υποψηφίου σε μέτα. Μπορείτε να μετάτε στη μητρική σας γλώσσα, διότι έχουμε διερμηνία σε 22 γλώσσες. Η συνεδρίαση αναμεταδίδεται μέσω του διαδικτύου. Είναι δημόσια. Και θα μπει μετά και στο δίκτυο του Κοινοβουλίου και τα πρακτικά το συντομότερο δυνατόν θα τα έχουμε και αυτά μετά τη συνεδρίαση. Το λόγο αμέσως στον ε, Επίτροπο Σεμέτα για μια εισαγωγή 10 λεπτών. Madame Monsieur le Κυρία Πρόεδρε, κύριε Κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αξιότιμοι βουλευτέ, Χαίρομαι ιδιαίτερα που βρίσκομαι σήμερα ενώπιον σα, ω υποψήφιο επίτροπο για την φορολογία εντελολυγιακή ένωση στον εσωτερικό έλεγχο και καταπολέμηση τη απάτη. Δηλαδή, ω υποψήφιο επίτροπο, που θα έχει στη διάθεσή του πάρα πολλά δημοσιονομικά μέσα και μέσα πληροφόρηση για να δημιουργήσει έναν κινητήρα με ένα μόνο καθήκον να οδηγεί στην Ευρώπη να μπορέσει να ανταποκριθεί στις προσδοκίες των λαών της. Η οικονομική πρόοδος, οι καλύτερες δουλειές και οι ισχυρότερες κοινωνικές εγγύησεις, αυτές είναι οι ελπίδες και ανάγκες των Ευρωπαίων σήμερα. Ασφάλεια από κακοβουλές ενέργειες και από ατυχήματα, η κλιματική αλλαγή, η ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος που έχουν όλα αυτά είναι ανησυχίες των Ευρωπαίων. Αυτές λοιπόν οι ελπίδες και οι ανησυχίες πρέπει να μας καθοδηγήσουν και θα αποτελέσουν το βασικό νήμα όλων μου των θα διατρέχει όλες μου τις ε, πράξεις. Βεβαίως η φορολογία είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα συλλογικό εισόδημα. Όπως επίσης και ο ιστορικός έλεγχος καταπολέμησης απάτης είναι κάτι περισσότερο από απλούς ελέγχους. Αυτά τα μέσα έχουν πολύ περισσότερες δυνατότητες, οι οποίες πρέπει να εκμεταλλευτούμε για να αναπτυχθεί οικονομικά και κοινωνικά η Ευρώπη. Εάν υποστηρίξετε λοιπόν την ε, υποψηφιότητά μου, θα γίνω μέλος της ε, Κομισιόν με ένα ευρύτατο χαρτοφυλάκιο που θα καλύπτει δύο τομείς, καθώς τα έσοδα και τα έξοδα είναι, αν θέλετε, δύο πτυχές του ίδιου κύκλου και πρέπει να έχουν τον ίδιο σκοπό, δηλαδή να έχουν το το για την κοινωνία. Και πρέπει να υπόκειται στις ίδιες αρχές διαφάνεια, απλότητα, λογοδοσία και υπευθυνότητα και βέβαιο σεβασμό για το χρήμα των φορολογουμένων. Είμαι πεπισμένος για όλα αυτά, οπότε η καταπολέμηση της οποιασδήποτε απάτης είτε έχει σχέση με τα έξοδα του προϋπολογισμού είτε με τους δασμούς είτε με τους φόρους θα είναι καθημερινό μου μέλημα. Δεν έχω καμία αμφιβολία πως όλα η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Καταπολέμησης Απάτης έχει πολύ σημαντικό ρόλο να παίξει εδώ πέρα κατά την ε, πρώτη δεκαετία έχει αποκτηθεί πάρα πολύ μεγάλη εμπειρία από τον Όλαφ και έχει αποκτήσει μια σημαντική φήμη. Εδώ πέρα λοιπόν θα ήθελα να αναφέρω τον Φραντς Χέρμαν Μπρίνερ, τον πρώτο γενικό διευθυντή του Όλαφ, ο οποίος δυστυχώς όπως ακούσατε απεβίωσε το κυριακό που μας πέρασε. Αλλά βεβαίως έχουμε όλοι τον ίδιο στόχο να επιτύχουμε μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, οπότε πρέπει να δούμε τα πράγματα μια νέα ματιά και να επιφέρουμε τις απαραίτητες αλλαγές. Ιδέες υπάρχουν, αλλά για να βρούμε την σωστή ιδέα θα πρέπει να είμαστε ανοιχτόμυαλοι, να εξερευνήσουμε όλες τις επιλογές, αυτές που είναι ήδη επιτάπητος και αυτές που θα αναπτυχθούν στο μέλλον. Η ανεξαρτησία του Όλαφ, οι διαφορετικές στοιχείες της λογοδοσίας του, το γραφείο του Ευρωπαϊκού Δημοσίου. Κατηγορού όλα αυτά είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Γνωρίζω λοιπόν πως έχεις αφήσει απόψη το Κοινοβούλιο εδώ πέρα, γι' αυτό σκοπεύω να τα συζητήσω όλα αυτά μαζί σας τώρα. Να περάσω στα... στην πλευρά των εξόδων του προπολογισμού. Μιλάμε για τα χρήματα του κόσμου. Δεν υπάρχει λοιπόν καμία δικαιολογία, τίποτα δεν μπορεί να δικαιολογήσει κατάχρηση αυτών των χρημάτων και αυτό ο έλεγχος θα αποτελέσει την πρώτη προτεραιότητα. Βεβαίω δεν ξεκινάμε από το μηδέν. Έχει υπάρξει σημαντική πρόοδο τα τελευταία χρόνια, όμως δεν πρέπει να σταματήσουμε τις προσπάθειές μας για να διασφαλίσουμε πώς θα υπάρχει, θα ξέρουμε πού πηγαίνει το κάθε ευρώ. Σκοπεύω επίσης να μειώσω το διοικητικό κόστος, ενώ ταυτόχρονα καταπολεμούμε τον διοικητικό κίνδυνο. Θα υπάρχει λοιπόν πλήρης ε, λογοσία εάν ε, κάποια κονδύλια διατίθενται είτε αχρεωστήτως είτε παρανόμως είτε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο. Οπότε δίνω μεγάλο βάρος και στην περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας της διαφάνειας. Επίσης, η ανάπτυξη συγκεκριμένων προτάσεων για το ανεκτό επίπεδο σφάλματος θα είναι ένα από τα βασικά μου καθήκοντα όσον αφορά τα έξοδα του προϋπολογισμού και είμαι θα συνεργαστούμε εδώ πέρα με τους συναδελφούς μου. Είναι απολύτως απαραίτητο να απλοποιηθούν οι κανόνες όσον αφορά τα κριτήρια επιλεξιμότητας ε, των ε, δικαιούχων των ευρωπαϊκών κονδυλίων και έτσι θα συντομεύσει η διαδρομή των χρημάτων αυτών προς τους δικαιούχους στα συγκεκριμένα έργα. Πιστεύω πως αυτό θα μας βοηθήσει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία μεταξύ της μεσονομικής φυταρχίας, της λογοδοσίας, της διαφάνειας και της άπλητας Και θεωρώ πως οι λύσεις αυτές ε, θα μπορέσουν να μας βοηθήσουν να προχωρήσουμε προς μια θετική ε, δήλωση διαβεβαίωσης και σε συνεργασία και με την ε, δική σα επιτροπή και με το ελεγκτικό συνέδριο θα προσπαθήσω να επιτύχω αυτούς τους στόχους. Θεωρώ πάρα πολύ σημαντική τη συνεισφορά σας και θα λάβω υπόψη αυτά τα οποία ακούστηκαν κατά τη διαδικασία απαλλαγής. Κυρίε και κύριοι βουλευτές, ως Υπουργός Οικονομικών και τους τελευταίους μήνες Επίτροπος Προϋπολογισμού έχω πλέον την πείρα θα έλεγα να αναλάβω αυτά τα καθήκοντα και θα έλεγα πως ε, έχω και μια ιδέα για τον αντίκτυπο που έχουν αυτά τα ποσά όχι μόνο σε εκατομμύρια στον προπολογισμό, αλλά το τι αποτέλεσμα έχουν στην κοινωνία, στην απασχόληση, στην κοινωνική ασφάλιση, στην οικονομική ανάπτυξη και μας δίνουν όλα αυτά τη δυνατότητα να κάνουμε αυτά τα οποία χρειάζεται η κοινωνία μας. Αυτή τη στιγμή η Ευρώπη βρίσκεται σε ένα κρίσιμο σημείο. Βγαίνουμε θα έλεγα από μια ελεύθερη πτώση όσον αφορά την οικονομία, όμως παραμένει εύθραυστη η κατάσταση, οπότε πρέπει να αναζωογονηθεί η οικονομία, αλλά και να έχουμε σταθερά δημοσιοοικονομικά. Οι φόροι πληρώνονται από τους πολίτες και οτιδήποτε κάνουμε επηρεάζει όλες τις οικογένειες στην Ευρώπη. Οπότε κάθε απόφαση πρέπει πρώτα απ' όλα να αντανακλά μια ιδέα, δεύτερον να αντικατοπτρίζει έναν δημόσιο στόχο και τρίτο και σημαντικότερο να συνεισφέρει στην εφαρμογή αυτών. Πώς λοιπόν θα τα επιτύχω αυτά στον τομέα της φορολογίας και των τελωνίων. Πρώτα απ' όλα θα δούμε τι θα γίνει με την εσωτερική αγορά, καθώς είναι οπωσδήποτε ένα από τα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά επιτεύγματα, αλλά πρέπει να ασκήσουμε και κάποια αυτοκριτική. Δεν εκμεταλλευόμαστε πλήρως τα πλεονεκτήματα της ε, εσωτερικής αγοράς. Πρέπει να δούμε ποια είναι τα φορολογικά εκείνα εμπόδια τα οποία δυσκολεύουν τους πολίτες και τις ε, επιχειρήσεις. Τέτοια φορολογικά εμπόδια πρέπει να καταργηθούν άμεσα. Όλα τα ζητήματα διπλής φορολογίας πρέπει να ε, επιλύονται γρήγορα και υπέρ των φορολογουμένων. Πρέπει να δούμε επίσης το τι θα γίνει με την κοινή φορολογητέα ύλη των ε, επιχειρήσεων. Θέλω να τονίσω αυτό, καθώς εάν έχουμε ένα ενιαίο τρόπο προσδιορισμού αυτής της φορολογητέας ύλης, θα έχουμε νέες ευκαιρίες στην εσωτερική αγορά, θα μειώσει το κόστος για τις εταιρείε, θα ευνοήσει την κινητικότητα και την ανταγωνιστικότητά μας. Επίσης, εντός και εκτός της Ένωσης ε, υπάρχει μείωση του διοικητικού κόστους, η απλοποίηση του φορολογικού συστήματος, ε, επίσης το να γίνονται πιο γρήγορα οι επιστροφές της εφορίας, ε, όλα αυτά τα ζητήματα μας απασχολούν. Επίσης ένα από τα πιο καυτά, αν μου επιτρέπετε, ζητήματα του καιρού μας είναι η ενέργεια. Σκοπεύω εγώ να προχωρήσω σε φορολογικές καινοτομίες για να ενισχυθεί η καινοτομία και η προστασία του περιβάλλοντος και θεωρώ πως πρέπει στην φιλοσοφία μας φορολογική να έχουμε μια έμφαση στα πράσινα ζητήματα. Επίσης θα εξυγχρονίσουμε τα τελωνία. Η Ευρώπη του 21ου αιώνα χρειάζεται ένα τελωνιακό σύστημα του 21ου αιώνα. Μιλάω εδώ πέρα για ηλεκτρονικά τελωνία που θα βασίζονται σε ένα σύγχρονο κώδικα και θα χρησιμοποιήσουν στο έπακρο την πληροφορική. Ένα τέτοιο τελωνιακό σύστημα θα χρησιμεύει και σε επιχειρήσει και στου πολίτε και θα εξοικονομεί χρόνο και χρήμα. Επιπλέον, μόνο αυτό το σύστημα θα μπορέσει να εκπληρώσει την αποστολή του δηλαδή να διασφαλίζει και τα σύνορά μας και τις αγορές μας και τα δικαιώματα της ε, πνευματικής ιδιοκτησίας και της ιδιοκτησίας γενικότερα. Ανέφερα λοιπόν συνεχώς ε, της προτεραιότητάς μου όσον αφορά την οικονομία και τον προπολογισμό και τη φορολογία, αλλά η οικονομία είναι ένα μέσο, δεν είναι αυτός σκοπός. Πρέπει να προωθεί φιλόδοξες ευρωπαϊκές ιδέες και να επιταχύνει τις αλλαγές που θέλουν οι άνθρωποι και να ενισχύσει ένα κοινωνικό μοντέλο στο οποίο κανείς δεν θα είναι στο περιθώριο. Είναι πολλά αυτά βεβαίως και θεωρώ πως ε, κλειδί για να επιτύχουμε είναι οι συντονισμένες προσπάθειες όλων των θεσμικών εργάνων. Γι' αυτό η στενή συνεργασία μαζί σας θα αποτελεί καθημερινό μου μέλημα. Θεωρώ πως η εμπιστοσύνη είναι προαπαιτούμενο για τη συνεργασία μας, γι' αυτό θα σας ε, ενημερώνω όχι μόνο για τις επιτυχίες και τα επιθέματα, αλλά και όλα τα, για όλα τα προβλήματα που θα αντιμετωπίζουμε και ελπίζω το πρώτο βήμα του διαλόγου μας να είναι η σημερινή ακρόαση. Ευχαριστώ. Eh, Ευχαριστούμε κύριε τον Επιτροπό και το λόγο στην κυρία Γκρέσλη για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επίτροπε. Αυτή τη στιγμή είναι στο κέντρο έλεγχος του προπολογισμού και θα ήθελα και εγώ να καταγραφεί στα πρακτικά ο σεβασμός μου για το έργο του κυρίου Μπρούνερ και βεβαίω έχουμε τώρα το ζήτημα της ακαθόδου θέσης ε, του Όλαφ. Έχουμε το πρόβλημα το ότι η Κομισιόν εδώ και 14 μήνες μπροκάρει την μεταρρύθμιση του Όλαφ. Εσείς σκοπεύετε να υποβάλλετε μέχρι το τέλος του το σχετικό έγγραφο εργασίας για να μπορέσει να συνεχιστεί αυτή η μεταρρύθμιση του Όλαφ. Γιατί φοβόμαστε ότι θα ξεκινήσει ξανά τα πράγματα από την αρχή η Κομισιόν με τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα. Θα πάμε πάλι πίσω στο πρόγραμμα. Ο Γενικός Διευθυντής του Όλαφ έχει επίσης μεγάλη ευθύνη για τις ε, ε, έρευνες, το δεύτερο μου ερώτημα, και θα διορίζετε διοργανικά. Είστε έτοιμος για τέτοιες διοργανικές λύσεις και υπενθυμίζω εδώ πέρα πως η ιδιαίτερη ευθύνη ε, που υπάρχει εδώ πέρα στο ε, Κοινοβούλιο είναι ακριβώς πως θα υπάρξει στην κεφαλή του Όλαφ ένας εισαγγελέα. Είστε διατεθειμένος να ακολουθήσετε μια τέτοια πορεία. Ευχαριστώ. Κομισάριο, Uh, uh, Ευχαριστώ. Θα ήθελα να αρχίσω από το δεύτερο ερώτημα και νομίζω ότι κοινό μας καθήκον είναι να εξασφαλίσουμε την συνέχεια των δραστηριοτήτων της Όλαφ. Και νομίζω ότι η Επιτροπή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να εξασφαλίσει αυτή τη συνέχεια ήρθαμε σε επαφή με τις νομικές υπηρεσίες για να βρούμε την κατάλληλη λύση επί του θέματος. Γνωρίζετε ότι ο κύριος Κάλλας είναι ακόμα υπεύθυνο για τις δραστηριότητες της Όλαφ και θα συνεργαστούμε μαζί του στενά επί του θέματος. Είμαι έτοιμος να συζητήσω μαζί σας όλους τους ενδεχόμενους τρόπους να προχωρήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι ο βασικός μας στόχος είναι να διασφαλίσουμε το συντομότερο δυνατόν την, τον διορισμό ενός νέου Γενικού Διευθυντή και αναμένω την πλήρη σας υποστήριξη και συνεργασία έτσι ώστε να βρούμε τον καταλληλότερο τρόπο ε, περιγραφής του έργου του νέου Γενικού Διευθυντή της Όλαφ σε σχέση με την νομοθεσία που διέπει την Όλαφ, νομίζω ότι είναι απαράδεκτο το γεγονός ότι η Επιτροπή δεν αντέδρασε στις προτάσεις του Συμβουλίου καθώς και τις προτάσεις του Κοινοβουλίου ως προς τη νομοθεσία αυτή η οποία υποβλήθηκε, πρόταση νομοθεσίας που υποβλήθηκε στο Κοινοβούλιο το 2006 και είχαμε τις δικές σας προτάσεις το Νοέμβριο του 2008 ως απάντηση. Ξέρετε τη δέσμευση του Προέδρου Μπαρόζο που εξέφρασε κατά τη διακήρυξη των Γενικών Κατευθυντηρίων Γραμμών ως προς την Όλαφ και η πρόταση αυτή υποστηρίχθηκε από μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, γι' αυτό θα βρούμε τους κατάλληλους τρόπους να βρεθεί μια τελική λύση. Κρέσλο για ένα λεπτό. Το γεγονός πως ε, στις ε, οδηγίες ε, του κυρίου Μπαρόζο αναφέρεται πως θα πάει προς μια εξωτερική υπεργολαβία το έργο του Όλοφ δεν νομίζω πως είναι πάρα πολύ θετικό. Εμείς ήμασταν πάντα ως κοινοβούλιο ΚΑ πώς σκοπεύετε να λύσετε αυτή την διαμάχη. Θέλετε να διατηρηθεί ο Όλαφ τμήμα της ε, Κομισιόν. Δεν αντιλήφθηκα την απάντησή σας. Επίσης το εάν θα υποβάλλετε το έγγραφο εργασίας για τη μεταρρύθμιση του Όλαφ ή όχι. Ευχαριστούμε πολύ. Ο Επίτροπος για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Το συζητήσαμε λεπτομερώς το θέμα αυτό με τον πρόεδρο Μπαρόζο και μπορώ να σας εγγυηθώ ότι ο Πρόεδρος προτίθεται να εφαρμόσει τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που υποστήριξε και η μεγάλη πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Θεωρεί λοιπόν ότι οι πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές δεν είναι απλώς ένα χαρτί, είναι πραγματικές κατευθυντήριες γραμμές που θα ήθελε να εφαρμόσει στην πράξη δηλαδή κατά τη μελλοντική του εργασία. Βεβαίως θα πρέπει να βρούμε τρόπους ε, για την αντιμετώπιση του ζητήματος και εδώ παραμένω ανοιχτό σε υποδείξεις δικές σας για να δούμε πώς μπορούμε να εξασφαλίσουμε το ανεξάρτητο και αποδοτικό καθώς και αποτελεσματικό έργο της Όλαφ. Ευχαριστώ. Γκέιερ για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε κύριε Επίτροπε, θα επανέλθω στον Όλαφ. Είναι επεποίθηση της Επιτροπής μας πως ε, ο Όλαφ ε, πρέπει να είναι όσο δυνατόν πιο αποτελεσματικός, καθώς η καταπολέμηση της απάτης αποτελεί βασικό αντικείμενο της πολιτικής μας και είμαστε πεπισμένοι πως η καταπολέμηση της απάτης είναι τομέας στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορεί να χαλαρώσει και το παρακολουθεί πάρα πολύ στενά η κοινή γνώμη αυτό το θέμα. Είπατε στην, ε, στις δηλώσεις ε, του Μπαρόσο πως ε, πράγματι αυτές έγιναν θετικά δεκτές από την πλειοψηφία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου πράγματι αλλά ξέρετε πως υπήρχε πάρα πολύ μεγάλη αποχή η δική μου ομάδα καταψήφισε και γνωρίζουμε ήδη τις πλειοψηφίες. Αν είναι να λέμε πως ε, υπάρχει ε, πλειοψηφία για κάτι, δεν ανάγκη να συνεδριάζει το, το Κοινοβούλιο. Θέλω να απαντήσετε εάν πράγματι θέλετε να παραμείνει ο Όλαφ κομμάτι της Κομισιόν. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Επαναλαμβάνω την πρώτη μου απάντηση ως προς το εξής. Ε, αυτό που είναι πολύ σημαντικό για την Όλαφ είναι να είναι ένα ανεξάρτητο και αποτελεσματικό σώμα. Μέχρι τώρα η Όλαφ ε, επετέλεσε αυτό το έργο για να καταπολεμήσει την απάτη και τη διαφθορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εδώ θα πρέπει να αποτίσουμε φόρο τιμή στον κύριο Μπρίνερ, τον πρώτο Γενικό Διευθυντή της Όλαφ. Θα πρέπει να συνεχίσουμε το ίδιο έργο με την ίδια διάθεση. Θα πρέπει να συνεργαστούμε για να εξεύρουμε τον καλύτερο δυνατό τρόπο να προωθήσουμε την τελική λύση για την Όλαφ, έτσι ώστε να είναι ένα ανεξάρτητο σώμα και να λάβουμε υπόψη και το θέμα της Ευρωπαϊκής Γενικής Εισαγγελίας. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να συνδυάσουμε αυτά τα δύο, τα δύο ζητήματα, πώς να βρούμε τον καλύτερο τρόπο λειτουργίας αυτού του θεσμού και αυτό αφορά και τον Ευρωπαίο Εισαγγελέα, Γενικό Εισαγγελέα. Αυτό το συζητήσαμε με την κυρία Ρέντινγκ, με την Πρωταθήσα Επίτροπο και είμαστε έτοιμοι να συνεργαστούμε μαζί της επί του θέματος αυτού. ένα λεπτό. Θεωρώ πως το ζήτημα της ανεξαρτησίας του Όλαφ δεν, δεν το συζητάμε. Αυτό το υποστηρίζουμε όλοι σε αυτή την Επιτροπή. Το ζήτημα είναι πώς θα εργαστεί πιο αποτελεσματικά εάν δεν είναι πλέον τμήμα της Κομισιόν αλλά ξεχωριστή υπηρεσία και θα είναι απ' έξω αν θέλετε από τον κοινοτικό μηχανισμό. Εάν κατάλαβα καλά τον ε, κύριο Μπαρόσο σκοπεύει να κάνει αυτόνομη οντότητα τον Όλαφ. Πώς κρίνεται, πώς θα διασφαλίσετε μάλλον την ε, αποτελεσματικότητα έτσι του Όλαφ έναντι των λοιπόν θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ο Επίτροπος για ένα λεπτό. Το ουσιώδες ζήτημα είναι η αποτελεσματικότητα, η αποδοτικότητα της εργασίας της Όλαφ. Νομίζω ότι οι πολίτες μας δεν ενδιαφέρονται για την ε, θεσμική ταυτοποίηση της Όλαφ. Αυτό που σε ενδιαφέρει περισσότερο είναι οι δραστηριότητες της Όλαφ για την καταπολέμηση της απάτης και της διαφθοράς καθώς και η αντιμετώπιση άλλων σοβαρών ζήτημάτων. Εδώ θα πρέπει να αξιολογήσουμε όλα τα υπέρ και τα κατά. Τι ακριβώς χρειάζεται για να εξασφαλίσουμε αυτό το έργο, έτσι ώστε να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες των πολιτών. Δέχομαι οποιαδήποτε πρόταση σε κάθε λεπτομέρεια για τη μελλοντική, για τη εξέλιξη του θεσμού αυτού, της Όλαφ. Ευχαριστούμε πολύ. Χατζημαρκάκης για ένα λεπτό. Κύριε Επίτροπε, εμείς εκπροσωπούμε τους πολίτες της Ευρώπης, γι' αυτό να σας πω και για την τρίτη ομάδα, πως είναι πρόβλημα το να βγει εκτός κομισιόν η Όλαφ είμαστε όλοι κατά. Να αναφέρω κάτι άλλο τώρα. Τι μη κυβερνητικέ οργανώσεις. Και εδώ πέρα υπάρχει απάτη ή μπορεί να υπάρξει απάτη και διαπιστώνουμε πω η Κομισιόν αρνείται μέχρι στιγμή να ορίσει τις ΜΚΟ και να μας δώσει μια σαφή εικόνα για το ποιε ΜΚΟ υποστηρίζει. Αυτά. Ενώ ορίζουν την πολιτική πολλών επιτρόπων και αναφέρω εδώ πέρα ε, προστασία καταναλωτών και κυρίως του περιβάλλοντος. Ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, ποιο τους έχει εκλέξει δημοκρατικά. Δεν υπάρχει λοιπόν προστασία, δεν υπάρχει διαφάνεια όσον αφορά το να ξεκαθαρίσει κομισιόν φορολογούμενους τι κάνουν τα χρήματά τους. Σκοπεύετε να ε, ελέγξετε την συμπεριφορά των ε, μη κυβερνητικών οργανώσεων όσον αφορά την κοινωνική του χρηματοδότηση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ Επίτροπος για να απαντήσει. Νομίζω ότι το, το ζήτημα των μη κυβερνητικών είναι πολύ σημαντικό. Είναι σοβαρότατο, συμφωνώ μαζί σας. Το θέμα του ορισμού, ως προς το πρόβλημα του ορισμού, νομίζω ότι αν μαζί μπορούμε να, μπορέσουμε να βρούμε μια κοινή περιγραφή των μη κυβερνητικών θα βοηθούσε ιδιαίτερα για την αντιμετώπιση του ζητήματος, να βρούμε κοινού ορισμούς δηλαδή. Συμφωνώ μαζί σας, αλλά το πρόβλημα έγκυται στο εξής. Εάν δούμε τις εθνικές νομοθεσίες που ορίζουν τις μη κυβερνητικέ, βλέπουμε ότι υπάρχει ε, μεγάλη ε, απόκληση και είναι δύσκολο να βρούμε έναν κοινό παρονομαστή για τον ορισμό των ε, μη κυβερνητικών αλλά νομίζω ότι θα ήταν ε, πολύ χρήσιμο να γίνει κάτι τέτοιο. Σε σχέση με τη διαφάνεια, νομίζω ότι πολλά καταφέραμε γιατί μέσω διαδικτύου ε, μπόρεσαν να καρποθούν από τα αποτελέσματα όλοι οι δικαιούχοι των ε, μη κυβερνητικών και μπορεί κανείς σήμερα να κοιτάξει στο διαδίκτυο να δει ποια χρήματα έχουν ε, κατανεμηθεί ή δοθεί οπουδήποτε. Νομίζω ότι το διαδίκτυο και οι πύλες του, οι ιστότοποι δείχνουν που, ποιοι είναι οι δικαιούχοι στα κράτη-μέλη. Βεβαίως δεν είναι ο καλύτερος δυνατός αυτός ο ιστότοπος, θα πρέπει να γίνει πιο φιλικός προς το χρήστη και να βρούμε τρόπους ε, να δημιουργήσουμε καλύτερες μηχανές αναζήτησης έτσι ώστε οι πολίτες να έχουν περισσότερες δυνατότητες. Αυτό αφορά και την Όλαφ για να δούμε τι συμβαίνει με τους δικαιούχους τάχιστα και όποτε χρειάζεται. Ο κύριο Χατζημαρκάκης για ένα λεπτό. Να υπενθυμίσω πω ε, αυτή τη φορά δεν είναι μόνο τα κράτη-μέλη που δεν έκαναν σωστά τη δουλειά του, αλλά ούτε και η Κομισιόν. Δεν κατάφερε να κάνει μία λίστα είτε σε site είτε γραπτό και να μα τη δώσει. Χαίρομαι για το ότι το συζητάτε αυτό μαζί μας. Θέλω να ρωτήσω, εάν είναι δυνατόν να έχουμε μια τέτοια ενιαία λίστα ή site ή οτιδήποτε, ε, τώρα και με την ε, νέα κατανομή των αρμοδιοτήτων των επιτρόπων. Θεωρείτε εσείς ε, πως ε, θα οδηγήσουν τα νέα χαρτοφυλάκια, καθώς ο κύριος Κάλλας πριν είχε ευρύτερες αρμοδιότητες, ε, στο να μην ξέρουμε πλέον ποιε είναι οι αρμοδιότητε των επιτρόπων και να μπορούν όλοι να κρύβονται πίσω από το σώμα των επιτρόπων συνολικά. Και τι σκοπεύετε να κάνετε για να μην συμβεί κάτι τέτοιο. Ένα λεπτό για την απάντηση. Μπορώ να σας πω από κατανοώ εγώ το ζήτημα, ότι όλες οι πληροφορίες για τους δικαιούχους κονδυλίων της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα πρέπει να αφορούν μία ε, διαφανή διαδικασία μεταξύ Κοινοβουλίου και πολιτών, διότι πρόκειται για τα χρήματα των φορολογουμένων. Και οι φορολογούμενοι μας, οι πολίτες μάλλον, πρέπει να γνωρίζουν πώς δαπανώνται αυτά τα χρήματα και από ποιο φορέα. Υπάρχουν λοιπόν ε, σφάλματα στο σύστημα. Οι ελληπείς πληροφορίες θα ήθελα να συνεργαστώ μαζί σας για να βρούμε την καλύτερη δυνατή λύση. σε ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, πίσω σας είμαι. Κύριε, κύριε Πιτροπά. από πίσω σας είμαι. Κύριε Επίτροπε. Είμαι ο μόνιμος ε, εισηγητής για τα ίδια μέσα αυτής της ε, Επιτροπής και ασχολούμαι ζητήματα ΦΠΑ, απάτης και λοιπόν ε, υπολογίζεται ξέρετε ο ΦΠΑ γύρω στα 600 δισεκατομμύρια το χρόνο, η ιδέα πάτη γύρω στα 200 δισεκατομμύρια έχουμε αναλάβει λοιπόν πρωτοβουλίες και έχουμε κάνει πάρα πολλές συστάσεις και όσον αφορά την ε, απάτη και όσον αφορά την απάτη στο τράνζιτ και όσον αφορά το λαθρεμπόριο τσιγάρων. Σκοπεύετε να λάβετε κάποια συγκεκριμένη προτεραιότητα να πείτε ότι αυτό το ζήτημα εγώ θα το αντιμετωπίσω τα επόμενα δύο μισή χρόνια. Ποια μέτρα σκοπεύετε να λάβετε συγκεκριμένα προτεραιότητα. Διάβασα τις ε, εκθέσεις σας με πολύ ενδιαφέρον και έχω διαβάσει και άλλες εκθέσεις από άλλους ευρωβουλευτές και τις βρίσκω πολύ ενδιαφέρουσες τις εκθέσεις αυτές. Μας δίνουν στοιχεία να σκεφτούμε τι μέτρα μπορούμε να λάβουμε Συμφωνώ με αυτό που είπατε, ότι η απάτη όσον αφορά το ΦΠΑ απαιτεί επιπλέον μέτρα. Η Επιτροπή ήδη έχει προτείνει πολλά μέτρα προς το Συμβούλιο. Καταρχήν να επιταχυνθεί η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών. για το ΦΠΑ στα εισαγόμενα που ήταν, από τα, ήταν ένα από τα παραθυράκια του συστήματος. Το Συμβούλιο ήδη έχει αποφασίσει γι' αυτό. Το ίδιο πρέπει να κάνουμε με την απάτη καρουσέλ, που είναι το πιο καυτό θέμα. Η Επιτροπή πρότεινε το διοικητικό σύστημα, το λεγόμενο Eurofisk. Νομίζω το σύστημα Eurofisk και η αποτελεσματική ανταλλαγή πληροφοριών για τις περιπτώσεις απάτης είναι τα δύο πιο σημαντικά θέματα. Πρόεδρος, ο κύριος Στάς, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Επιτροπέ πρέπει να πω πως ε, συχνά μιλάμε για εγκληματικά δίκτυα και πολύ δημιουργικά όσον αφορά την απάτη καρουσέλ. Μόλις την προηγούμενη εβδομάδα στο Βέλγιο συνελήφθησαν δύο Βρετανοί υπήκοοι γιατί ήταν ε, αναμεμειγμένοι σε εμπόριο καρουσέλ δικαιωμάτων εκπομπών. Δηλαδή μιλάμε σε πάρα πολύ διαφορετικά αντικείμενα ε, όταν μιλάμε για καρουσέλ ε, στον ΦΠΑ των δικαιωμάτων εκπομπών είναι πολύ σοβαρά τα πράγματα. Και διαβάζουμε εδώ πέρα πάρα πολύ συχνά τις εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου και δεν νομίζω ότι παίρνουμε αρκετά σοβαρά αυτά τα πράγματα και πρέπει να δούμε όντως να δοθεί κάποια συνέχεια αυτό. Θα ήθελα λοιπόν να σας παρακαλέσω να κάνετε κάποιο σχόλιο. Ε, Διάβασε την έκθεση του ελεκτικού συνεδρίου και τις συστάσεις. Πρέπει να τις λάβουμε υπόψη μας. Αυτές οι συστάσεις πρέπει να εφαρμοστούν από την Επιτροπή. και αυτό θα είναι προτεραιότητα για μένα στη μελλοντική μου δουλειά. Για τις απάτες για το ΦΠΑ θα μπορούσε να συνεργαστεί και η Όλαφ με την δραστηριότητα αυτή. Βέβαια για θέματα φορολόγησης τα περισσότερα εμπόδια βρίσκονται στα κράτη-μέλη. Και πρέπει να δούμε βέβαια και τι πόρους διαθέτει ο Όλαφ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Έπινγκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ερώτηση. Τι θα κάνετε με τις ειδικές εκθέσεις του ελεγκτικού συνεδρίου, ιδιαίτερα στην περιφερειακή πολιτική και την ανάπτυξη. Μερικέ φορέ δεν υπάρχουν λεφτά, μερικέ φορέ τα λεφτά δεν δαπανώνται με σωστό τρόπο ή δεν πετυχαίνουμε του στόχου. Ένα συγκεκριμένο παράδειγμα σε σχέση με την ερώτηση Χατζημαρκάκη για την ε, πολιτική ανάπτυξη. Πέρυσι ένα δι δαπανήθηκαν από μη κυβερνητικέ οργανώσει. και τα περισσότερα από τα χρήματα αυτά δεν δαπανήθηκαν σωστά. Το επικρίνει το Ελληνικτικό συνέδριο. Πολλά προγράμματα δεν είναι καν βιώσιμο που είναι πολύ σημαντικό για τέτοιου είδους προγράμματα. Και ένας έχει 50.000 προγράμματα, πολλά από τα οποία δηλαδή και ιδιαίτερα στο τομέα των διαρθρωτικών ταμείων. Και για το 2008 βλέπουμε ότι το ποσοστό σφάλματος είναι της τάξης του 11%. Αυτό είναι απαράδεκτο από κάθε άποψη, γι' αυτό θα πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια αντιμετώπισης των δαπανών στον τομέα των διαρθρωτικών ταμείων. Από την άλλη πλευρά όμως θα πρέπει να υπάρχει μια σαφής ε, διαφορά μεταξύ σφαλμάτων και απάτης διότι η πλειονότητα των σφαλμάτων ε, σχετίζονται με την έλλειψη τεκμηρίωσης και την ε, παραβίαση των ε, κριτηρίων εκλεγιμότητας ή άλλα ζητήματα, ας το πούμε ίσονος σημασίας, αλλά η απάτη είναι το μείζον ζήτημα και ξέρετε ότι υπάρχουν παραδείγματα αναστολής πληρωμών και ανέκυψαν και περιπτώσεις με την Βουλγαρία και τη Ρουμανία στο παρελθόν, τέτοιες περιπτώσεις. Γι' αυτό η Επιτροπή ελέγχει τα συστήματα εποπτείας των κρατών μελών και είναι έτοιμη να αναλάβει δράση εκεί όπου χρειάζεται. Ζώντερ ένα λεπτό. Ευχαριστώ και ήλπιζα να απαντήσει με ένα ναι απλά ο κύριος Επίτροπος, το οποίο δεν το έκανε. Θα ήθελα να γνωρίζω εάν εσείς προσωπικά σκοπεύετε να δεσμευτείτε ότι δεν θα δοθούν πλέον κονδύλια στις χώρες και στις περιφέρειες εκείνες οι οποίες γίνεται συνεχώς κακοδιαχείριση των χρημάτων. Και κάτι ακόμα, το οποίο επίσης μπορείτε να απαντήσετε με ένα ναι ή με ένα όχι. Συμφωνείτε μία φορά το έτος να έρχεστε ενώπιον της Επιτροπής μας και να ξεκαθαρίσετε τυχόν αντικρουόμενα συμφέροντα εντός της Κομισιόν. Παραδείγματο χάρη στην ε, τελευταία Επιτροπή Μπαρόζου υπήρχαν πάρα πολλά συγκρουόμενα συμφέροντα. Υπήρχε επίτροπος ο οποίος είχε επιχειρήσεις, άλλος ο οποίος ήταν σύμβουλος της ε, Microsoft ε, και ταυτόχρονα σύμβουλος ε, επιτρόπου. Θα έρχεστε εδώ πέρα για να ξεκαθαρίζετε τέτοια συγκρουόμενα συμφέροντα. Remember. Απάντηση. Κύριε Βούλευτα, νομίζω ότι η Επιτροπή αναλαμβάνει κάθε δράση που χρειάζεται όταν υπάρχουν αποδείξεις απάτης ή σφαλμάτων. Υπάρχει ένα σύστημα ε, χρηματοπιστωτικών επανορθώσεων και το 2008 το επίπεδο επανόρθωσης ανήλθε σε 3 δις ευρώ. Και η αναστολή πληρωμών χρησιμοποιήθηκε και 10 φορές ε, το 2008 σε σχέση με το 2007 που χρησιμοποιήθηκε μόνο μία φορά. Βλέπετε λοιπόν ότι επιτελούμε αυτή την εργασία καλώς, αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι θα πρέπει να καταβάλουμε μεγαλύτερες προσπάθειες σε αυτό το τομέα, έτσι ώστε να βελτιώσουμε ακόμα περισσότερο την πλαισίωση αυτή στα κράτη-μέλη και ως προς τη σύγκρουση συμφερόντων, ναι, βεβαίως μπορώ να προσέρχομαι στο Κοινοβούλιο και να συζητώ οποιοδήποτε θέμα ανακύπτει στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ. Αντρέσεν για ένα λεπτό. Thank you, Chairman. Mr. Semeta. Ευχαριστώ. Κύριε Σεμέτα, στην απάντησή σας στο ερωτηματολόγιο μιλήσατε πάρα πολύ θετικά για τον θεσμό του Ευρωπαίου Εισαγγελέα θα επιμείνετε στην ε, σύσταση ενός ε, τέτοιου θεσμού παρά το βέτο το οποίο προβλέπεται από την πολιτική κυβέρνηση κατόπιν. Ε, τι γίνεται με τον νέο κώδικα συμπεριφοράς των επιτρόπων. Τρίτο ερώτημα. Γνωρίζετε πως ο Γενικός Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου αυτή τη στιγμή ήταν ο αρχιλογιστής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Δεν βλέπετε κάποιο πρόβλημα με το να ελέγχει, τουλάχιστον για τα δύο πρώτα χρόνια, το ίδιο του το έργο αυτός ο άνθρωπος. Και τέταρτο ερώτημα. Υπάρχουν πάρα πολλές συζητήσεις κάθε φορά που δημοσιεύουν οι ελεγκτές την έκθεσή του για σφάλματα ή απάτες. Ποιος είναι ο δικός ορισμός της απάτης. Ευχαριστώ δύο λεπτά για την απάντηση. Για το ζήτημα του εισαγγελέα. Είναι δύσκολο ζήτημα. Είχαμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση συζητήσεις ε, πολλές ε, για αυτό το ζήτημα το, το 2000-2001, αλλά νομίζω πως ε, η συνθήκη της Λισαβόνας επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Ένωση να συστήσει ένα τέτοιο αξίωμα μπορούμε να, πρέπει να κυριθούμε προς αυτήν την κατεύθυνση και όπως ανέφερα και στην αρχή συζητήσαμε αυτό το ζήτημα με την ε, κυρία Ρέντινγκ και θα συνεργαστούμε από αυτού. Η άποψή μου είναι πως ε, ένα γραφείο τέτοιο του Ευρωπαϊκού Εισαγγελέα θα βοηθήσει να αποτελεσματικότερη λειτουργία της Ένωσης όσον αφορά τον κώδικα συμπεριφοράς των επιτρόπων. είναι πολύ σημαντικό να προχωρήσουμε σε αυτόν τον τομέα. Ο κύριος Μπαρόσο το ανέφερε αυτό στις κατευθυντήριες γραμμές του. Οπότε η Κομισιόν ε, θα είναι έτοιμη να συνεργαστεί με σας και με το Συμβούλιο σε διοργανικό επίπεδο και είναι νομίζω πολύ σημαντικό να αυξηθεί το πώς ε, να γίνει πιο γνωστός ο κώδικας συμπεριφοράς. Ε, γι' αυτό θα πρέπει να συνεργαστεί διοργανικά η Κομισιόν με το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και να συζητήσει την δυνατότητα να αποτελέσει ένα υπόδειγμα αυτός ο κώδικας για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό νομίζω. Ε, ίσως μια ερώτηση μου ξέφυγε, η τελευταία ερώτηση για το Γενικό Διευθυντή. Σας ε, Αντριάσεν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας έλεγα ότι ο γενικό Διευθυντής ήταν ο πρώην επίτροπος, ο κύριος ε, Chief Accountant δεν θεωρείτε ότι υπάρχει σύγκρουση εδώ συμφερόντων σε σχέση με τα δύο τελευταία χρόνια. Είναι σαν να ελέγχει κατά κάποιο τρόπο τον εαυτό του. Απάντηση. Ο Μπράιον Γκρέι είναι ένας πολύ συνετός άνθρωπος και συζητήσαμε το θέμα των δραστηριοτήτων στην υπηρεσία γενικού ελέγχου, General Audit. Έχει πάρα πολλές ιδέες σχετικά το πώς μπορεί να βελτιωθεί η λειτουργία της υπηρεσίας εσωτερικών ελέγχων. Και όσον αφορά τη σύγκρουση, ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων, ορίζεται στον ε, εσωτερικό κανονισμό. Στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν νομίζω ότι υπάρχει τέτοια περίπτωση σύγκρουση συμφερόντων. Έρεν Άουζερ, e- ένα λεπτό. Απουσιάζει κάποιο άλλο από του μη εγγεγραμμένους. Θέλει να μιλήσει στη θέση του. κανεί. Προχωρούμε. Οντί, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Στην δήλωση διαπίστευση. ο πρόεδρος Μπαρόσο έδωσε θετικό ντάς εκ μέρου του Ελληνικού Συνεδρίου και έχουμε πολύ λίγα στοιχεία στην μία δήλωση του κυρίου Μπαρόσο. Βέβαια έχουμε και την γραπτή σα απάντηση και ρωτώ η αλυσίδα ελέγχου, η ποιότητα, ιδιαίτερα στην κοινή διαχείριση με τα κράτη-μέλη. Ποια είναι η άποψή σας. Δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να συμπεριλάβουμε και τα εθνικά ελεγκτικά συνέδρια, το επιτρέπουν οι συνθήκες, και τα εθνικά κοινοβούλια, για να έχουμε κοινή δουλειά, γιατί ο ρόλος του κοινοβουλίου είναι να ελέγχουν την εκτελεστική εξουσία. Εμά ο ρόλος μας είναι να ελέγχουμε την Επιτροπή. Δεν θεωρείται για να έχουμε καλή ποιότητα ελέγχων το ανεκτό περιθώριο λάθος κλπ. να έχουμε μια καλύτερη ποιότητα στην αλυσίδα ελέγχου. Πρόεδρος, δύο λεπτά για την απάντηση. Ναι. Θεωρώ ότι κι άλλη δουλειά για τα θετικά DAS και μάλιστα πιο ενεργή δραστηριότητα απαιτείται και μπορούμε να το πετύχουμε αν συνεργαζόμαστε. προκειμένου να λυθούν θέματα που σχετίζονται με διάφορα παρεθυράκια που υπάρχουν στο σύστημα. Ξέρετε ότι το κύριο πρόβλημα στις δαπάνες είναι η δαπάνη κοινοτικών κονδυλίων σε εθνικό επίπεδο. Τώρα έχουμε ένα νέο σύστημα αιτήσεων συνοπτικών καταστάσεων για δύο χρόνια. Η ποιότητα των αιτήσεων αυτών καταστάσεων, annual summaries, δεν είναι ακόμα ικανοποιητική. Έχουμε και την πρόταση για το δημοσιονομικό κανονισμό με τροπολογίες. Αυτό θα ενισχύσει τον ε, έλεγχο όσον αφορά το δημοσιονομικό κανονισμό και τα, η θετική δήλωση αξιοπιστίας είναι τμήμα των απαιτήσεων. και τα ελεγκτικά όργανα θα μπορούν να φέρουν σε πέρας πιο εύκολα το έργο τους. Βέβαια, εδώ υπάρχει το θέμα της επικορικότητας. Πρόεδρος, ο συνάδελφος Οντί, δευτερολογία ένα λεπτό. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Ένα λεπτό, ο κύριος Σταυρακάκης. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ κύριε Υποψήφιο Επίτροπε, στις γραπτές σας απαντήσεις τονίζετε ως προτεραιότητα καλή ποιότητα ε, δημοσιονομικής δαπάνης με περισσότερη διαφάνεια, λιγότερη γραφειοκρατία, περισσότερο αίσθημα ευθύνη και υπολογία. Όσον αφορά την κακοδιαχείριση, και απολύτω συμφωνώ με όλα αυτά. Αν λάβουμε υπόψη όλα αυτά, πώ θα βελτιώσετε τα συστήματα ελέγχου των πόρων τη Ένωση, ώστε οι δικαιούχοι τη πολιτική συνοχή, ιδιαίτερα μικρέ οργανώσει, μικρέ τοπικέ αρχέ, μη κυβερνητικέ οργανώσει και άλλοι κοινωνικοί εταίροι, να έχουν πιο εύκολη πρόσβαση στα κονδύλια αυτά με υγιή διαχείριση και με λιγότερα ποσοστά λάθος. Πρόεδρος, η απάντηση δύο λεπτά. Φύγεται ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Ξέρετε, τα τελευταία χρόνια Έχουμε φτάσει σιγά σιγά στην τελική φάση διαχείρισης των συστημάτων ελέγχου στα κράτη-μέλη και η Επιτροπή θεωρεί ότι το νέο σύστημα θα επιτρέψει καλύτερο έλεγχο των συστημάτων που ισχύουν στα κράτη-μέλη. Η ερώτησή σας, αν την κατάλαβα καλά, αφορά την απλοποίηση των κανόνων. Συμφωνώ με τα πορίσματα του ελεγκτικού συνεδρίου και αυτή είναι η προσωπική μου γνώμη ότι υπάρχει κι άλλο περιθώριο απλοποίησης των κανόνων σχετικά με τις δαπάνες. Γιατί όσο πιο πολύπλοκοι οι κανόνες, τόσο πιο μεγάλη η δυνατότητα, μάλλον η πιθανότητα λαθών. Έχουμε μια καλή ευκαιρία τώρα, διότι ο δημοσιονομικός κανονισμός υφίσταται αναθεώρηση, έχει ξεκινήσει μια δημόσια διαδικασία διαβούλευσης για τον κανονισμό από τον Οκτώβριο. Έχουμε πάρει μερικές καλές προτάσεις για βελτίωση του δημοσιονομικού κανονισμού Έχουμε και εμείς τις δικές μας ιδέες και το Ευρωκοινοβούλιο έχει αυτό μερικές ωραίες ιδέες. Πιστεύω ότι θα καταλήξουμε σε προτάσεις που θα οδηγήσουν σε σημαντική απλοποίηση του δημοσιονομικού κανονισμού που θα μας επιτρέψουν να έχουμε πιο εύκολη ε, δαπάνη, πιο εύκολη για τους δικαιούχους με υγιή ε, δημοσιονομική διαχείριση ταυτόχρονα. Πρόεδρος, ε, έχετε ένα λεπτό για να δευτερολογήσετε. Ευχαριστώ, δεν έχω άλλο σχόλιο κύριε Πρόεδρε. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Και τώρα ένα λεπτό, Μάρκο Μπέι, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Στην περιγραφή του χαρτοφυλακίου σας αναφέρεται ο κ. Μπαρόζο στην καταπολέμηση της απάτης ε, και της φοροδιαφυγής. Όπως ξέρουμε, οι φορολογικοί παράδοση χρησιμοποιούνται και από Ευρωπαίους επιχειρηματίες για να αποφύγει την ευρωπαϊκή φορολόγηση το εισόδημά τους. Το ερώτημα, τι συγκεκριμένα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για να σταματήσει αυτή η φόρο διαφυγή και οι παράνομες δραστηριότητες ε, των ε, υπεράκτιων φορολογικών παραδείσων. Είναι, έχετε ως προτεραιότητα κάτι τέτοιο. Ποιο είναι το χρονοδιάγραμμά σας και κάτι σχετικό. Δεσμεύεστε να ξαναξεκινήσετε την διαδικασία έγκρισης της ε, οδηγίας περί προστασίας από το ποινικό δίκαιο των συμφερόντων της κοινότητας το οποίο μπλόκαρε το Συμβούλιο το 2001 και του κανονισμού για την ε, αμοιβαία διοικητική αρρωγή για την ε, προστασία των συμφερόντων της κοινότητας που επίσης μπλόκαρε το Συμβούλιο και τον μπλοκάρει από το 2004. Σας ευχαριστώ δύο λεπτά. Ναι. Νομίζω πως ε, το ζήτημα των φορολογικών αυτών παραδείσων. Είναι κρίσιμο αυτή τη στιγμή όταν τα κράτη-μέλη αντιμετωπίζουν ε, σημαντικές ε, δυσκολίες. Και γνωρίζετε πως λόγω της κρίσης ε, το επίπεδο του χρέους των κρατών μελών αυξάνεται. Και πρέπει να καταβάλουμε κάθε προσπάθεια έτσι ώστε να υπάρξει ορθή διοίκηση και διακυβέρνηση στο σύστημα της ε, φορολογίας και έχουν γίνει αρκετά πράγματα. Ήδη γνωρίζετε πως η Επιτροπή διαπραγματεύεται μια συμφωνία με το Λιχτενστάιν, ε, μια συμφωνία καταπολέμησης απάτης και εάν ε, καταλήξουμε σε συμφωνία θα αποτελήσει αυτή πρότυπο και για άλλα ευρωπαϊκά κράτη όπως η Ανδόρα, το Μονακό, το Σαν Μαρίνο και η Ελβετία. Και νομίζω πως ε, επίσης ε, η οδηγία και η σχετική συζήτηση για τις καταθέσεις είναι πάρα πολύ κρίσιμη και νομίζω πως θα καταλήξουμε σε μια λύση και θα πείσουμε τα υπόλοιπα δύο κράτη-μέλη που μπλοκάρουν ε, την οδηγία μαζί με ένα πακέτο άλλων οδηγιών στο οποίο πακέτο περιέχεται και αυτή η οδηγία αμοιβαίας αρρωγής. Και βεβαίως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε κάθε μέσο που έχουμε, ειδικά της αναπτυξιακής συνεργασίας ε, και να ε, ενσωματώσουμε, να θέσουμε το ζήτημα της ε, σωστής ε, διακυβέρνησης, στις διαπραγματεύσεις μας ε, με τους εταίρους μας ε, για την αναπτυξιακή συνεργασία για να διασφαλίσουμε πως η ορθή διακυβέρνηση θα αποτελέσει αρχή των φορολογικών συστημάτων και εντός της Ένωσης και στον υπόλοιπο κόσμο. Οπότε αυτό αποτελεί προτεραιότητά μου και θα ασχοληθώ πάρα πολύ με αυτό. Για την άλλη οδηγία θα τη μελετήσω προσεχώς. Και αν μια νέα πρόταση οδηγίας ε, είναι να αυξήσει την αποτελεσματικότητα, οπωσδήποτε θα κινήσω την διαδικασία. Μακοβέ για ένα λεπτό. Είπατε πώς υποστηρίζετε την αναθεώρηση του υπάρχοντος κώδικα συμπεριφοράς. Σκοπεύετε λοιπόν να ασχοληθείτε με τα κενά, όπως το ότι δεν υπάρχει σαφής ορισμός των αντικρουόμενων συμφερόντων, το ότι δεν υπάρχει σαφήνεια όσον αφορά τα δώρα, και να συμπεριληφθεί και η φιλοξενία, όπως οι προσκλήσεις για διακοπές σε αυτή την κατηγορία. Η έλλειψη σαφών κριτηρίων για το πώς ορίζεται η συμβατότητα για απασχόληση μετά την θητεία, ε, ναι ή όχι, σας παρακαλώ, και σκοπεύετε να ευθύσετε τον νέο κώδικα συμπεριφοράς μέχρι τον Ιούνιο 2010. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό. Όπως ε, ανέφερα, η Επιτροπή θα επεξεργαστεί τον ε, νέο κώδικα συμπεριφοράς και θα προσκαλέσει όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα και το Κοινοβούλιο δηλαδή να βοηθήσουν σε μια διοργανική ομάδα εργασίας ε, για να καταθέσεις κατάλληλες προτάσεις. Από τα ζητήματα τα οποία αναφέρατε, πράγματι ε, είναι ζητήματα που πρέπει να μας απασχολήσουν, αλλά πρέπει να δούμε τον κώδικα συμπεριφοράς σε ένα ευρύτερο πλαίσιο συζητήσαμε με τον ε, πρόεδρο τον κύριο Μπαρόσο πως ο κώδικας αυτός συμπεριφοράς θα αποτελέσει πρότυπο για όλα τα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα για να έχουμε σωστή συμπεριφορά όλων των ε, θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό, σαλτεμόζε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ως ε, βουλευτές είμαστε εκπρόσωποι των Ευρωπαίων πολιτών και βεβαίως ε, θέλουμε να γνωρίζουμε το τι γίνεται σε όλες τις δραστηριότητες της ε, Ένωσης και στα έξοδα. Εσείς τι, ε, πώς το βλέπετε, το δικαίωμά μας δηλαδή να μπορούμε να έχουμε άποψη και να βλέπουμε και τι γίνεται με τη διαδικασία απαλλαγής. Σας ευχαριστώ δύο λεπτά. Η άποψή μου είναι πολύ απλή. Νομίζω ότι οι βουλευτές έχουν κάθε δικαίωμα ελέγχου των δαπανών η κάθε δαπάνη από πλευράς ευρωπαϊκού προϋπολογισμού και νομίζω ότι οι προηγούμενες διαδικασίες απαλλαγής καταδεικνύουν ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει επιτελέσει μια πολύ σοβαρή εργασία και πολύ καλές συστάσεις. για την πιο αποτελεσματική διαχείριση των κοινοτικών πόρων. Το 2007 είχαμε 203 συστάσεις από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και η Επιτροπή εφήρμοσε τις 195 από αυτές. Νομίζω λοιπόν ότι αυτό είναι ο καλός τρόπος εξασφάλισης της αποτελεσματικότητας της δαπάνησης των κοινωτικών κονδύλιων. Θα συνεχίσω αυτή την αποτελεσματική εργασία μαζί σας με βάση τις συστάσεις σας, τις οποίες θα προσπαθήσω να εφαρμόσω. Δεν υπάρχει άλλη ερώτηση. Δελάνς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε, εγώ το ότι έκανα προεκλογική εκστρατεία για να βγω αποδεικνύει και το ότι έτρεξα με συγχωρείτε για να μπω στην αίθουσα αποδεικνύει το ότι θέλω να σας κάνω πραγματικά πάρα πολύ ερώτηση. Ξέρετε πως ε, είναι πάρα πολύ μεγάλη προτεραιότητα μας η διαβεβαίωση, η θετική διαβεβαίωση. Ήταν η Κομισιόν στο πλευρό μας. Βλέπουμε πως οι συνόψεις αυτές δεν έχουν μεγάλη προσθέμενη αξία. Από το ερώτημά μου είναι εσείς ως υποψήφιος και ως επίτροπος τι σκοπεύετε να κάνετε έτσι ώστε οι δηλώσεις να γίνουν ετήσιες ε, δηλώσεις διαχείρισης και ε, μπορούμε να βασιστούμε επάνω σας ως Κοινοβούλιο και Επιτροπή για να μας υποστηρίξετε σε αυτό το πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα στην επόμενη διοργανική συμφωνία και τις δημοσιονομικές προοπτικές. Ευχαριστώ. Δύο λεπτά για την απάντηση. Αυτό το ζήτημα ε, αφορά εγγυήσεις δαπάνης των ε, κοινοτικών πόρων. Αυτό το θέμα είναι ύψη τη σημασία και δεν υπάρχει καμία αμφιβολία, δεν χωρεί αμφιβολία. Ξέρετε ότι προσπαθήσαμε ως Επιτροπή να ορίσουμε ένα σύστημα εθνικών δηλώσεων διαχείρισης το 2005, αλλά η πρόταση αυτή απορρίφθηκε από το Συμβούλιο. Και ανταυτής ε, προτάθηκαν ε, ετήσιες ε, ανακεφαλαιώσεις ε, οι οποίες έγιναν αποδεκτές αλλά με ορισμένες δυσκολίες από το Ευρωπαϊκό, Κοινοβούλιο, ε, Συμβούλιο. Με συγχωρείτε. Όπως ήδη προανέφερα, μέσα στα πλαίσια της δήλωσης αξιοπιστίας θα θέλαμε να προωθήσουμε αυτές τις διασφαλίσεις και ήδη 11 κράτη-μέλη το προέβαλαν και τέσσερα κράτη-μέλη ε, προβάλλουν μια ετήσια δήλωση καθώς και δήλωση αξιοπιστίας για το 2008. Άρα συνολικά έχουμε 11 κράτη-μέλη που υποβάλλουν δήλωση αξιοπιστίας, άρα γνωρίζουμε πώς δαπανώνται οι πόροι. Στα πλαίσια της αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού θα πρέπει να προχωρήσουμε περαιτέρω έτσι ώστε να έχουμε μια καλύτερη περιγραφή και απαιτήσει για τα κράτη-μέλη. Τουλάχιστον θα πρέπει να έχουμε εθελούσιες ετήσιες δηλώσεις διαχείρισης. Το έχω συζητήσει με τα κράτη-μέλη το ζήτημα αυτό, διότι εμπλέκονται άμεσα τα κράτη-μέλη και αυτό που έχει σημασία είναι η εργασία που διέπει είτε τις αιτήσιε συγκεφαλαιώσεις είτε τις αιτήσιε δηλώσεις διαχείρισης. Και νομίζω ότι εδώ μπορεί να επιτελεστεί πρόοδος και βελτιώσει. Ένα λεπτό. Δεν χρειάζομαι ένα λεπτό, αλλά εγώ σας ρώτησα πώς. Πώς ε, και ποιες πρωτοβουλίες θα αναλάβετε. Έχετε ένα περιθώριο ελιγμό, αλλά τι θα κάνετε έμπρακτα. Εξ αρχής ανέφερα ότι βρισκόμαστε τις ενώπιον της διαδικασίας αναθεώρησης του δημοσιονομικού κανονισμού και η Επιτροπή θα υποβάλει μια πρόταση το Μάιο του 2010 για την αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού και αυτά, αυτό θα είναι ένα από τα πρώτα βήματα έτσι ώστε να έχουμε νέες ιδέες στον ε, δημοσιονομικό κανονισμό σε σχέση με τις ετήσιες δηλώσεις ή τις ετήσιες ε, δηλώσεις διαχείρισης. Μετά, ο κανονισμός θα υποβληθεί στο Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο και θα συζητήσουμε την πρόταση αναθεώρησης ε, επινώντας την καλύτερη δυνατή λύση και για τα δύο θεσμικά όργανα. Γκέρπραντ, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντελάνγκε υπέβαλε το ίδιο ερώτημα με αυτό που θα ήθελα να υποβάλω κι εγώ. Αλλά δεν με ικανοποίησε η απάντησή σας. Γι' αυτό θα επεκταθώ. Αν κατανόησα καλά, πιστεύετε στη διαφάνεια και πιστεύω ότι η διαφάνεια είναι το μόνο μέσον για να έχουμε ένα καλύτερο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα ε, διαφάνειας και δαπάνης του δημόσιου χρήματος βρίσκεται στα έγκυται στα κράτη-μέλη. Άρα δεν αρκεί να είμαστε πιο ανοιχτοί στον τρόπο διαχείρισης. Θα πρέπει να επιβάλλουμε στα κράτη-μέλη να μας δώσουν ετήσιες δηλώσεις και ετήσιες ανακεφαλαιώσεις για το πώς θα πανούν τα χρήματα αυτά. Άρα θα επινοήσετε μια νέα πρόταση έτσι ώστε τα κράτη-μέλη να υποβάλουν ετήσιες δηλώσεις. Θα πρέπει να είμαστε ιδιαίτερα αυστηροί από αυτού. Απάντηση για δύο λεπτά. για να απαντήσω στο, μάλλον απαντώντας στο προηγούμενο ερώτημα, ανέφερα ότι τάσομαι υπέρ των εθνικών δηλώσεων διαχείρισης, αλλά θα πρέπει να είμαστε ρεαλιστές ως προς αυτή την απόφαση, διότι ξέρετε ότι η απόφαση για τον δημοσιονομικό κανονισμό θα ληφθεί στα πλαίσια συναπόφασης ε, δυνάμει της συνθήκης της Λισαβόνας. Ως προς τις ε, επί του προϋπολογισμού αρχές, δηλαδή του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Άρα θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξεύρουμε την καλύτερη δυνατή λύση. Στην προηγούμενη μου απάντηση τόνισα ότι αυτό που έχει μεγάλη σημασία είναι η εργασία που, που διέπει αυτή την προετοιμασία είτε των ετησίων συγκεφαλαιώσεων είτε των ετησίων δηλώσεων. Και αυτή την άποψη συμμερίζεται και το ελεγκτικό συνέδριο. Διότι αν δεν υπάρχει ε, επαρκής ποιότητα στη προγενέστερη εργασία, τότε θα έχουμε απλώς ένα κομμάτι χαρτί και τίποτα άλλο. Θα πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι γίνονται οι σωστοί έλεγχοι από τη, τα εθνικά θεσμικά όργανα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα έτσι ώστε να έχουμε πλήρη εξασφάλιση του γεγονότος ότι οι δηλώσεις είναι πραγματικές δηλώσεις αξιοπιστίας και βασίζονται σε ευρήματα σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα. Αυτό είναι ύψης της σημασίας. Ε, για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ για αυτή την απάντηση, αλλά γνωρίζετε όπως και εγώ ότι στα πλαίσια του Συμβουλίου υπάρχει αρχή του μη παρεμβατισμού σε σχέση με τη δαπάνη ευρωπαϊκών κονδυλίων στα κράτη-μέλη. Είναι προς δικό του συμφέρον, να μην υπάρχει παρεμβατισμός, γιατί έτσι ο καθένας μπορεί να ταπανεί τα χρήματα όπως ορίζει. Ε, εάν λοιπόν ε, μπείτε στα χωράφια του Συμβουλίου δεν θα φτάσουμε πουθενά. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, θέλετε να δώσετε μάχη προς αυτή την κατεύθυνση, δηλαδή να προβάλλετε μεγαλύτερη διαφάνεια από τα κράτη-μέλη για τον τρόπο δαπάνησης του δημοσίου χρήματος. Το να μας λέτε θα το κάνουμε από κοινού δεν αρκεί. Πρόκειται για μια μεγάλη μάχη που θα πρέπει να δώσετε και δεν ξέρω κατά πόσο θέλετε να συμπαραταχθούμε σε αυτό το τομέα. Ευχαριστώ. Ένα λεπτό για την απάντηση. Είμαι υπέρ των αποτελεσμάτων, των απτών αποτελεσμάτων. Και αυτό που έχει μεγάλη σημασία για μένα είναι η επίτευξη ενός αποτελέσματος με βάση τις στοχοθετήσεις μας. Και νομίζω λοιπόν ότι θα πρέπει να συνεργαστούμε με τα κράτη-μέλη έτσι ώστε να εξεύρουμε μια λύση που θα μας επιτρέψει να βελτιώσουμε την αποτελεσματικότητα της δαπάνησης των κοινοτικών κονδυλίων και αυτό είναι αναπόσπαστο μέρος του, των καθηκόντων μου. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το επίπεδο σφάλματος είναι απαράδεκτο. Από την άλλη πλευρά πιστεύω ότι τα νέα συστήματα που ήδη επιβάλλονται για τη νέα περίοδο προγραμματισμού γιατί θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι το ελεγκτικό συνέδριο εκπώνησε εκθέσεις με βάση το παλαιό ε, δημοσιονομικό πλαίσιο Τώρα υπάρχει και η μίνιντας, η μικρή δήλωση αξιοπιστίας, έτσι ώστε να μειωθεί το περιθώριο σφάλματος. Άρα κινούμαστε προς την ε, σωστή κατεύθυνση και, αυτές είναι και, αυτή είναι και η πρόθεσή μου. για ένα λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε, παρατηρούμε στην συζήτηση βεβαίως πως έχετε δύσκολο χαρτοφυλάκιο και έχετε να ασχοληθείτε και με το Συμβούλιο. Θα ήθελα όμως εγώ να αναφερθώ στο συλλογικό όργανο. Έχετε ένα οριζόντιο χαρτοφυλάκιο, γι' αυτό θα πρέπει να ε, έρθετε σε επαφή και με τους λοιπούς επιτρόπους, με τα λοιπά χαρτοφυλάκια και να τους πείστε να κινηθούν με πλήρη διαφάνεια έναντι του Κοινοβουλίου. Με ποια συγκεκριμένα σας παρακαλώ μέτρα θα φροντίσετε για να υπάρξει πρόοδος στα προβληματικά χαρτοφυλάκια και συγκεκριμένα πώς σκοπεύετε να διασφαλίσετε την λεπτομερή συνολική εικόνα των λοιπόν χαρτοφυλακίων για να εφαρμοστούν συγκεκριμένα αυτά τα οποία έχει ζητήσει το Κοινοβούλιο κατά τη διαδικασία της απαλλαγής. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ δύο λεπτά. Yes, I... Ναι, συμφωνώ. Ε, είναι σημαντικό να ορίσουμε μια γενική διαδικασία στην Επιτροπή έτσι ώστε οι συστάσεις και τα ευρήματα των διαφόρων αρχών να εφαρμόζονται σωστά. Θεωρώ ότι τα τελευταία χρόνια η Κομισιόν σημείωσε σημαντική πρόοδο σε αυτό. Χρειαζόμαστε συγκεκριμένα εργαλεία για να αντιμετωπίσουμε τα θέματα που αναφέρατε. Έχουμε επιτροπή πρόοδου του ελέγχου, στην οποία θα προεδρεύω στο μέλλον. Και αυτή η Audit Progress Committee, αυτή η επιτροπή πρόοδου των ελέγχων, θα βοηθήσει σε βελτιωμένη δράση της Κομισιόν. Βέβαια πρέπει να συντονιστεί ακόμα καλύτερα η δραστηριότητα αυτής της ε, Επιτροπής ιδιαίτερα σε περιοχές υψηλού κινδύνου πρέπει να ενισχυθεί το σύστημα διαχείρισης του κινδύνου στην Επιτροπή και η Επιτροπή αυτή πρόοδο των ελέγχων, όπως σας είπα, να εστιαστεί στους υψηλούς κινδύνους. Αυτό αποτελεί τμήμα των υποχρεώσεών μου. Είναι της ευθύνης μου στους γενικούς ελέγχους όπως επίσης και ο καλύτερος συντονισμός της Επιτροπής αυτής και η εστίαση της δραστηριότητάς της σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Πρόεδρος, η κυρία Ολμέγερ έχει και ένα ακόμη λεπτό αν θέλει. Να επανέλθω. Πώς βλέπετε τη συνεργασία με τον Όλαφ. Συγκεκριμένα, Θα ήθελα δηλαδή να δω πώς θα συνενοηθείτε μαζί τους να, να κάνουν ό,τι λέτε. Και δεύτερον, πώς βλέπετε τις ε, προσπάθειες του Κοινοβουλίου για να έχει μία συνυπευθυνότητα στο μέλλον όσον αφορά την απαλλαγή και για την βελτίωση της ε, αξιοπιστίας και των δηλώσεων αξιοπιστίας. Uh, Yes, I think that's... Uh, για την Όλαφ αυτή τη στιγμή έχουμε όργανα που δεν αποτελούν κομμάτι της Κομισιόν Η Επίτροπη είναι αρμόδιοι για την συνεργασία και τον συντονισμό της δράσης αυτών των υπηρεσιών. θα πρέπει να βρούμε τον σωστό τρόπο για στενή συνεργασία μεταξύ της Επιτροπής και της ΟΛΑΦ. Πρέπει να δούμε το νομικό πλαίσιο. για σαφείς ε, διαφανείς τις ευθύνες της ΟΛΕΦ, της Επιτροπής και της συνεργασίας. Αυτό όμως είναι ένα πιο μακρόπνο σχέδιο και δουλειά. Πρόεδρος. Μπάλς για ένα λεπτό. Μπαλέστης. Κύριε υποψήφιο επίτροπε, μιλήσαμε αρκετά για την Όλαφ. Η υπηρεσία καταπολέμησης απάτης. Ωστόσο, εκθέσεις της Όλαφ μας λένε ότι πολύ συχνά διάφοροι θεσμοί και όργανα, που παραδείγματος χάρη υπεύθυνα για την εφαρμογή του νόμου στα κράτη-μέλη, καθυστερούν στο να εφαρμόσουν τις συστάσεις της Όλαφ όσον αφορά τις απάτες και την φοροδιαφυγή. Και ρωτώ, τι μέτρα θα λάβετε έτσι ώστε να λειτουργούν πιο υπεύθυνα όλα αυτά τα όργανα και οι θεσμοί. Δύο λεπτά απάντηση. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω στη μητρική μου γλώσσα. Συμφωνώ με αυτό που είπατε ότι τα πορίσματα των ελέγχων της ε, Όλαφ και η συνέχεια που δίνεται στις συστάσεις είναι ανεπαρκή. Πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι οι νομικές διαδικασίες συνήθως παίρνουν πολύ χρόνο και είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε συγκεκριμένα συμπεράσματα μετά από δραστηριότητα ενός ή δύο ετών μόνο. Προετοιμαζόμενος για την ακρόαση, μελέτησα διαδικασίες που κράτησαν μέχρι και 15 χρόνια. Τελικά, πετύχαμε αυτά αποτελέσματα. Ασκήθηκε δίωξη δηλαδή αυτών οι οποίοι επιδίδονταν σε δραστηριότητες απάτης. Πιστεύω ότι η κατάσταση μπορεί να βελτιωθεί. Υπάρχουν προτάσεις και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, από την κυρία Γκρέσλε συγκεκριμένα, για τρόπους βελτίωσης της συνεργασίας μεταξύ εθνικών οργάνων που φροντίζουν για την εφαρμογή της νομοθεσίας και των αντίστοιχων ευρωπαϊκών. Η εφαρμογή του νόμου βέβαια είναι ένα εθνικό θέμα. Αλλά η ανταλλαγή πληροφοριών και η υποβολή πληροφοριών σχετικά με τις διαδικασίες οι οποίες έχει κινήσει η Όλαφ, τις φάσεις σε οποίες βρίσκονται οι διάφορες διαδικασίες αυτές, όλα αυτά θα διευκολύνουν την καλή λειτουργία του συστήματος. Ευχαριστώ, Πρόεδρος. Δευτερολογία ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε υποψήφιο επίτροπε. Στην εισαγωγή σας μας ε, αναφέρατε ένα σημαντικό μελλοντικό έργο που είναι η απλοποίηση του συστήματος φορολογίας για κάθε κράτος μέλος. Μπορείτε σύντομα να μας πείτε τι έχετε κατά νου. Ένα λεπτό κύριε Σεμέτα. Λιθανικά. Το φορολογικό σύστημα απαιτεί αξιολόγηση της κατάστασης. Και μην ξεχνάμε ότι πρέπει να έχουμε υπόψη μας πάντα και την αρχή της επικορικότητας, που σημαίνει ότι όλες οι αποφάσεις σε θέματα φορολογίας παίρνονται ομόφωνα, με ομοφωνία επαναλαμβάνω στο Συμβούλιο. Ωστόσο υπάρχουν τομείς που μπορεί να γίνει απλοποίηση παραδείγματος χάρη σε θέματα κοινωνικού εμπορίου, ανταλλαγής πληροφοριών, θέματα διπλής φορολόγησης. Για αυτά τα θέματα σκοπεύουμε να κινήσουμε δημόσια διαβούλευση σε όλη την Ένωση, να εντοπιστούν τα εμπόδια σχετικά με την διπλή φορολογία και τα πιο επίγοντα προβλήματα και για τους επιχειρηματίες και για τους πολίτες. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τα προβλήματα αυτά. Μετά έχουμε το θέμα του ΦΠΑ. Οι πρωτοβουλίες που έχουν ήδη ξεκινήσει θα μας, βελτιώσουν, θα μας βοηθήσουν να βελτιώσουμε την κατάσταση. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Ήταλα, ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Μία ερώτηση για τα διορθωτικά ταμεία. 11% του κόστους στα διορθωτικά ταμεία ε, είναι παρατυπίες. Έχουν γίνει ένα σωρό έλεγχοι. Προσπάθησαν άκτηση των κονδυλίων με, ε, με μικρό αποτέλεσμα και το πρόγραμμα δράσης δεν βελτίωσε ιδιαίτερα την κατάσταση. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Μας μιλήσατε για τη δυνατότητα κυρώσεων αν οι συνθήκες δεν σας ικανοποιούν. Αλλά οι κυρώσεις αυτές δεν απέδωσαν στην περίπτωση ανάκτησης των κονδυλίων. Τι σκοπεύετε να κάνετε. Απάντηση. Δύο λεπτά. Συμφωνώ με αυτό που λέτε ότι το επίπεδο σφάλματος 11% δεν είναι ικανοποιητικό και πρέπει να το αντιμετωπίσουμε. Φυσικά πρέπει να λάβουμε υπόψη μας ότι η έλεγχη του ελεκτικού συνεδρίου είναι αιτήσιοι. Ενώ η Επιτροπή λειτουργεί ένα πολιετές σύστημα διαχείρισης και ελέγχου. Ένα παράδειγμα. Μόλις τώρα έκλεισε η περίοδος 94-99 και το υπολοιπόμενο περιθώριο σφάλματος είναι 3% για την περίοδο αυτή, 94-99. Εδώ δεν έχουμε και πολλούς τρόπους να βελτιώσουμε την κατάσταση. Τι έχουμε. Όσον αφορά την απλοποίηση καταρχήν. Πολλά σφάλματα δημιουργούνται γιατί οι κανόνες είναι πολύ πλοκοί. Και η Επιτροπή ήδη πρότεινε το 2009 ιδέες για την απλοποίηση και η αναθεώρηση του δημοσιονομικού κανονισμού θα μας ε, βοηθήσει να προχωρήσουμε αρκετά. Αυτό το είπε και το ελεγκτικό συνέδριο. Εντόπισε τα σημαντικά εμπόδια όσον αφορά την χρήση των διαρθρωτικών κονδυλίων. Η έννοια του ανεκτού ποσοστού σφάλματος είναι μια άλλη πρωτοβουλία θα την προτείνω και το 2010 η Επιτροπή θα κάνει συγκεκριμένες προτάσεις και μετά το θέμα του ποιος είναι υπόλογος. Η βελτίωση των αιτήσεων συνόψεων και των ε, αιτήσεων ε, δηλώσεων αξιοπιστίας, όλα αυτά θα βοηθήσουν το σκέλος του ποιος και πόσο είναι υπόλογος. Ήταλα, δευτερολογία ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ τον υποψήφιο για την απάντηση. Έχουμε ένα πρόβλημα επειδή δεν υπάρχουν δείκτες, κριτήρια γενικά αποδεκτά προκειμένου να μετρηθεί το πώς χρησιμοποιούνται τα δημόσια κονδύλια. Πιο γενικά, ερωτώ, έχουν γίνει αρκετά για να μετρηθεί η αξιοπιστία, η αποδοτικότητα μάλλον των κοινωτικών προγραμμάτων και πώς μπορούμε να αναπτύξουμε τέτοιου είδους κριτήρια. Απάντηση ένα λεπτό. Συμφωνώ. Μέχρι στιγμής κυρίως έχουμε ασχοληθεί με το αν επιλέξουμε μια δαπάνη με το ποσοστό ασφάλματος η δική μου άποψη είναι ότι πρέπει να οριστεί το ποσοστό σφάλματος. Είναι απαράδεκτο να έχουμε υψηλό ποσοστό σφάλματος σε συγκεκριμένες δαπάνες. Αλλά αυτό δεν αρκεί πρέπει να περάσουμε στην μέτρηση της αποδοτικής χρήσης των κονδυλίων. Άρα χρειαζόμαστε παραμέτρους και δείκτες. Δείκτες απόδοσης. Στο προηγούμενο έργο μου στη, στη Λιθουανία ασχολήθηκα με τα θέματα αυτά. Είναι ιδιαίτερης ιδιάζουσας σημασίας και είναι μια από τις σημαντικές μελλοντικές δραστηριότητες της Νέας Επιτροπής. Πρόεδρος, Herzog, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Εδώ στα αριστερά σημεία, κύριε Επιτροπέ. Πρόσφατα συστάθηκαν πολλές εκτελεστικές αποκεντρωμένες υπηρεσίε. Ανησυχείτε για το ότι με αυτόν τον τρόπο γίνεται σχεδόν αδύνατη η εγγύηση του δημοσιονομικού ελέγχου μπορείτε να μας πείτε ποια μέτρα θα λάβετε για να υπάρξει στις αποκεντρωμένες υπηρεσίες έλεγχος. Ποιο σχέδιο έχετε. Δύο λεπτά. Για να απαντήσω γενικά, προσωπικά πιστεύω πως ε, το να βγει εκτός της ε, Κομισιόν, το να βγουν εκτός της Κομισιόν οι δαπάνες πρέπει να γίνεται μόνο στις περιπτώσεις στις οποίες ε, βελτιώνεται η αποτελεσματικότητα όσον αφορά τις εκτελεστικές αυτές ε, υπηρεσίες. Νομίζω πως υπήρξε μια πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου για το ότι οι δαπάνες και η σύσταση αυτών των υπηρεσιών σε συγκεκριμένες, ε, συγκεκριμένες τομείς βελτίωσε την αποτελεσματικότητα των δαπανών. Όταν λοιπόν γίνεται κάτι τέτοιο μπορούμε να προχωρήσουμε σε σύσταση τέτοιων ε, υπηρεσιών. Νομίζω πως έχουμε σοβαρότερα προβλήματα με τις λεγόμενες παραδοσιακές ε, ας πούμε, υπηρεσίες, ε, τις οποίες έχουμε αρκετές και όταν έχουμε εκτελεστικές υπηρεσίες υπάρχουν σαφείς ε, κανόνες και τυποποίηση της ε, οργάνωσής τους. Ενώ ε, στον τομέα των παραδοσιακών αποκεντρωμένων υπηρεσιών δεν συμβαίνει κάτι τέτοιο και τώρα έχουμε μια διοργανική ομάδα εργασία που ασχολείται με αυτό. Και θα παρουσιάσει στο προσεχές μέλλον προτάσεις για το πώς θα έχουμε κοινά πρότυπα για τις παραδοσιακές ε, αποκεντρωμένες υπηρεσίε για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Και ξέρετε πως όσον αφορά τις παραδοσιακές ε, αυτές υπηρεσίες η Κομισιόν έχει αναλάβει σαφείς δεσμεύσεις να μην δημιουργήσει νέες τέτοιες υπηρεσίες, αλλά υπάρχουν ε, και έκτακτες περιστάσεις όπως η τρέχουσα κρίση που μας αναγκάζει να κάνουμε συγκεκριμένες προτάσεις στον ε, χρηματοοικονομικό τομέα. Σας ευχαριστώ. Άλλο ένα λεπτό, κύριε Χέρτσοκ. Ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, αυτό ήταν το ερώτημά μου. Είπατε πως έχουμε βελτιωμένη αποτελεσματικότητα. Ποια μέτρα θα λάβετε για να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα. Δεν το βλέπω εγώ και έχουμε πολλά προβλήματα στην Επιτροπή Ελέγχου του Προπολογισμού όσον αφορά την αποτελεσματικότητα ακριβώ και ελπίζω να συνεργαστούμε σε αυτό τον τομέα. Σας ευχαριστώ. Παρακαλώ. Θα γνωρίζετε ίσως ε, πως η υπηρεσία εσωτερικού ελέγχου ελέγχει τις περισσότερες από τις αποκεντρωμένες υπηρεσίες και υπάρχουν κάποιες καλές προτάσεις που έγιναν ε, κατά το πρόσφατο παρελθόν και μία από τις προτάσεις που είναι επιτάπητος είναι να δούμε την δυνατότητα σύστασης μιας επιτροπής εσωτερικού ελέγχου που θα αναλύσει τις προτάσεις και θα υποβάλει συστάσεις ε, στην διοίκηση των ε, αποκεντρωμένων ε, αυτών υπηρεσιών για το πώς θα βελτιωθεί ο Αυτό γίνεται και στον ιδιωτικό τομέα. Βεβαίως μπορεί να υπάρξει μια κοινή τέτοια επιτροπή, διοργανική, νομίζω πως μπορούμε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Σας ευχαριστώ Λάμπερτς για ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, θα ήθελα και εγώ να ακολουθήσω τους φορολογικούς παραδείσους. Κάθε χρόνο η απάτη 250 δις το χρόνο και για να μην μιλήσουμε για την φόρο διαφυγή. Μια κατάφορη αδικία έναν των φορολογμένων που πληρώνουν του και είναι πήγον το θέμα γιατί η δημόσια οικονομικά είναι κρίση σε όλε τι χώρε μα. Με διαφέρει λοιπόν οι προτάσει σα για του φορολογικού παραδείσου που κρύβονται μέσα στα σύνδρα τη Ένωση. Συχνά ο φορολογικό ανταγωνισμό παίρνει τη μορφή νόμιμων μεθόδων όπω το Βέλγιο, την πατρίδα μου, που είναι φορολογική παράδειση. Δηλαδή, εσείς ως Επίτροπος για θέματα φορολογίας, πώς σκοπεύετε να καταπολεμήσετε αυτή τη μορφή φορολογικών παραδείσεων, φορολογικού ανταγωνισμού που επαναλαμβάνω προξενεί ζημιά στο γενικό συμφέρον. Απάντηση δύο λεπτά. I fully agree that uh, the... Συμφωνώ ότι το θέμα των φορολογικών παραδείσων είναι κρίσιμα σημασίας, ιδιαίτερα σήμερα στην οικονομική κρίση που περνάμε. Είμαστε στη φάση ε, συμφωνίας, συμφωνιών μάλλον για την καταπολέμηση της ε, απάτης, φορολογικής απάτης με το Liechtenstein. Έχουμε ακόμα μερικές λεπτομέρειες να συζητήσουμε και υπάρχουν και μερικές χώρες που ακόμα χωρισμένοι εννοώ, που δεν συμφωνούν με το πακέτο αυτό μέτρων κατά της απάτης. Άρα θα ασκήσουμε όση πίεση μπορούμε για να προχωρήσουμε. Η συμφωνία αυτή με το Λίχτενστάιν θα μπορεί να αποτελέσει βάση για παρόμοιες συμφωνίες με άλλες χώρες στην Ευρώπη. Ανδόρα, Μονακό, Άγιος Μαρίνος, Ελβετία. Βέβαια, η Επιτροπή χρειάζεται εντολή διαπραγματευτική για όλες αυτές τις συμφωνίες. Με την υπογραφή αυτών των συμφωνιών θα έχουμε πρόοδο. Παράλληλα, υπάρχουν προδιαγραφές του ΩΣΑ για ανταλλαγή πληροφοριών. Και ξέρετε ότι στην Ένωση εφαρμόζουμε την αρχή της αυτόματης ανταλλαγής πληροφοριών με εξαίρεση μερικών κρατών μερών που είχαν μια μεταβατική περίοδο. Αλλά έχουμε σωστή ανταλλαγή πληροφοριών. μεταξύ των χωρών της Ένωσης, μάλλον χωρών που είναι στην Ευρώπη αλλά δεν είναι μέλη της Ένωσης και των κρατών μελών, είναι ύψης της σημασίας προκειμένου να έχουμε χρηστή διαχείριση και λιγότερη φοροδιαφυγή και φοροαπάτες. Λάμπερτς για ένα λεπτό. Δεν απαντήσατε στο ερώτημά μου, κύριε Επίτροπε, διότι ε, μίλησα για φορολογικούς παραδείσους στα 27, στα 27 κράτη-μέλη. Πιστεύετε ότι αυτό θα πρέπει να είναι ο κανόνας και όχι η εξαίρεση. Ε, επίσης, ε, μιλήσατε για το γεγονός ότι είσαστε result-oriented, δηλαδή υπέρ των αποτελεσμάτων πρωτίστως. Άρα, αν ε, δεν συμφωνήσουμε σε επίπεδο 27, τότε θα πρέπει να προωθήσουμε την ενισχυμένη συνεργασία. Ευχαριστώ. Απάντηση για ένα λεπτό, σε ένα λεπτό. Ίσως ε, δεν κατανόησα το πρώτο σας ερώτημα περί φορολογικών παραδείσων, γι' αυτό ζητώ συγγνώμη. Αλλά όταν μιλάμε ε, για θέματα φορολογικού ανταγωνισμού εδώ, η θέση μου είναι απόλυτα σαφής τάσσομαι υπέρ του δίκαιου φορολογικού ανταγωνισμού, γιατί νομίζω ότι βοηθά και στην ε, ανάπτυξη της οικονομίας, αλλά θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την αθέμητη φορολογική, τον αθέμητο φορολογικό ανταγωνισμό και εδώ ε, έχουμε μία ομάδα για έναν κώδικα συμπεριφοράς έτσι ώστε να μην δεχτούμε τις ε, κακές πρακτικές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει να ενισχύσουμε αυτή τη δραστηριότητα σε σχέση με την ενισχυμένη συνεργασία τώρα. Πιστεύω ότι όταν διαπιστώνουμε ότι κάτι τέτοιο βοηθά την ενίσχυση της εσωτερικής αγοράς της Ευρωπαϊκής Ένωσης, θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε βάσει αυτών των δυνατοτήτων που προβλέπονται και από τη Συνθήκη της Λισαβόνας. Ευχαριστούμε. Πόκρος για ένα λεπτό. Εκτός μικροφώνου. Ο μιλητής. Sorry. So 2010 should have been the... Το 2010 θα έπρεπε εμείς να είμαστε η πιο ανταγωνιστική ε, περιοχή του κόσμου. Αποτύχαμε ε, δραματικά. Ο Χωσέ Λουίς Ροντρίγκες Σαπατέρο ανέφερε ότι το 2020 θα πρέπει να είναι η νέα προθεσμία. Ποια ειδικά μέτρα θα πρέπει να ληφθούν σε φορολογικό επίπεδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να είσαστε σαφείς, διότι αναφερθήκατε σε ορισμένους τομείς όπου προσυπογράφεται τον φορολογικό ανταγωνισμό. Σε άλλους τομείς θέλετε φορολογική εναρμόνιση. Γι' αυτό θα θέλαμε να μας πείτε ε, ποιου συγκεκριμένους φορολογικούς ε, τομείς θα πρέπει να καλύψετε, δηλαδή τις φοροαπαλλαγές ή άλλους τομείς. Επίσης, ε, πώς αποτιμά την εργασία του προκατόχου σας, του κυρίου Λάσλο Κόβατς. Δύο λεπτά για την απάντηση. Σας ευχαριστώ για την ερώτηση. Θα αρχίσω με το δεύτερο ερώτημά σας. Ο Λάσλο Κόβατς επιτέλεσε ένα πολύ καλό έργο στην Επιτροπή κατά την ε, θητεία Μπαρόζο 1. Πολλές προτάσεις υποβλήθηκαν προς το Συμβούλιο επί όλων των θεμάτων που σχετίζονται, που άπτονται του φορολογικού. Βεβαίως δεν είναι εύκολο να επιτευχθεί μία συμφωνία διότι προαπαιτείται ομοφωνία. Και γι' αυτό θα πρέπει να πείσουμε τα κράτη-μέλη ότι μία απόφαση ε, είναι απαιτούμενη μια απόφαση σε επίπεδο ευρωπαϊκό, κάτι καθόλου εύκολο. Τώρα, σε σχέση με συγκεκριμένες προτάσεις, πιστεύω ότι κατά τα επόμενα έτη θα πρέπει να δώσουμε τελική ε, μορφή στην εργασία μας ως προς το κοινό φορολογικό πλαίσιο, διότι είναι πολύ σημαντικό για τις επιχειρήσεις και θα ήθελα να δούμε και τον τομέα των υπηρεσιών, ιδιαίτερα ως προς τις ΜΜΕ, διότι οι ε, ΜΜΕ αντιμετωπίζουν πρόβλημα μέσα στα πλαίσια του CCCTB και θα έπρεπε να κινηθούμε προς αυτή την κατεύθυνση. Νομίζω ότι η οδηγία για την φορολόγηση της ενέργειας είναι ύψης της σημασίας και θα πρέπει να ε, λάβουμε μία απόφαση διότι το παρόν σύστημα εκπομπών καλύπτει το 50% των συνολικών ε, εκπομπών. Γι' αυτό θα πρέπει να θεωρηθεί ως ένα πρώτο βήμα προς την πράσινη φορολόγηση. Αν προχωρήσουμε με την πράσινη φορολόγηση και ε, μειώσουμε το κόστος της ΜΜΕ, τότε θα έχουμε βοηθήσει ιδιαίτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, Μπόκρος για ένα λεπτό. Αν το θεωρείς σκόπιμο, ευχαριστώ. Ας εστιάσουμε την προσοχή μας σε κάτι πιο συγκεκριμένο. Δηλαδή, διαφωνείτε με τον Γκέρχαρτ Σρέντερ, τον πρώην καγκελάριο που ήθελε να προβάλλει κυρώσεις στη Σλοβακία όταν είχε ε, ένα εφάπαξ, μια εφάπαξ φορολόγηση σε όλους τους τομείς και έτσι αυτό οδήγησε άλλες χώρες σε μια φορολογική μεταρρύθμιση. Άρα χρειαζόμαστε περισσότερο παρά λιγότερο, περισσότερη παρά λιγότερη φορολόγηση στο μέλλον αν θέλουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας. Ένα λεπτό για την απάντηση. Το, ο ορισμός του συστήματος είτε πρόκειται για, ένα, για μια ε, FAPAX φορολόγηση ή ένα άλλο σύστημα φορολόγηση, αυτό είναι εναπόκειται στα κράτη-μέλη. Αυτό που θα πρέπει να επιτύχουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο είναι να έχουμε καλύτερο συντονισμό μεταξύ κρατών μελών σε θέματα φορολόγησης αλλά όχι να αναλάβουμε όλες τις ευθύνες που αφορούν τα κράτη-μέλη. Διότι τα κράτη-μέλη είναι εκείνα που αποφασίζουν για τα έσοδα και τις δαπάνες, ποιες θα είναι οι κοινωνικές δαπάνες και ούτω καθεξής. Ε, εγώ προτίθεμαι να διοργανώσω ένα φόρουμ υψηλού επίπεδου για την φορολόγηση στα κράτη-μέλη με επικεφαλής τους υπουργούς των κρατών μελών για να μιλήσουμε για την ε, μελλοντική ε, εξέλιξη του φορολογικού συστήματος. Θα πρέπει να γίνουν πολιτικές συζητήσεις και πολιτικής συζητήσεις βάθος μεταξύ κρατών μελών. Τώρα ε, αναθέτω την, την ε, Προεδρία στην ε, Πρόεδρο Σάρον Μπούλς της ΕΚΟΝ και θα ήθελα να τηρήσετε τα, τις χρονικές προθεσμίες όπως κάναμε μέχρι τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Τα γνωστά ισχύουν. Το πρώτο ερώτημα εκ μέρους του ΕΛΚΑ από την κυρία Κράτσα. Δεν ξέρω που κάθεστε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, στις ε, γραπτές απαντήσεις σας υποστηρίζετε ότι πρέπει να επανεξετάσουμε τη σκοπιμότητα υιοθέτησης μιας κοινή ενοποιημένης φορολογικής βάσης για τις εταιρείες, CCCTB, αναφερθήκατε και σήμερα, Ήθελα να σας ρωτήσω ποια άλλα μέτρα σκοπεύετε να λάβετε για την αντιμετώπιση των φαινομένων φορολογικού ντάμπινγκ εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, ήδη αναφερθήκατε ότι είναι πολύ δύσκολο ε, να πιστούν τα κράτη-μέλη για την αντιμετώπιση του φαινομένου αυτού. Έχετε, θα πάρετε κάποιες πολιτικές πρωτοβουλίες. Ήθελα να ρωτήσω ποια είναι η βασική σας επιχειρηματολογία για να πείστε τα κράτη-μέλη προς αυτή την κατεύθυνση και να ρωτήσω πώς κρίνεται και την ε, μέχρι τώρα εφαρμογή του κώδικα δεοντολογίας για την αντιμετώπιση αυτών των επιζήμιων πρακτικών του φορολογικού ανταγωνισμού ε, και εν ώψη της σχετικής έκθεσης που εκπώνησε ομάδα εργασίας κατά τη διάρκεια της Σουηδικής Προεδρίας. Ευχαριστώ. Η απάντησή σας κύριε Σας ευχαριστώ. Νομίζω πως ε, ο δίκαιος ε, ανταγωνισμός στον τομέα της φορολογίας είναι κάτι που μας βοηθάει στο να προχωρήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχετε δίκιο στο ότι τα προηγούμενα έτη είχαμε δει κάποια μείωση του ύψους φορολογίας, ειδικά όσον αφορά τις επιχειρήσεις. Ναι, αν δούμε γενικά το επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από τη δεκαετία του 1990 πέσαν οι φορολογικοί συντελεστές κατά 12% περίπου, αν δεν κάνω λάθος αλλά ταυτόχρονα, εάν δούμε τα έσοδα, σε σχέση με το ΑΕΠ, είναι πάρα πολύ σταθερά. Οπότε στο επίπεδο των κρατών μελών τα κράτη-μέλη τα οποία μειώνουν τον συντελεστή διευρύνει τη φορολογική τους βάση, οπότε έτσι αντισταθμίζεται η μείωση των εσόδων λόγω της μείωσης του συντελεστή. Αλλά βεβαίως υπάρχουν και κάποιες επιβλαβείς ε, πρακτικές που πρέπει να καταπολεμηθούν και υπάρχουν νέες εξελίξεις ε, όπως ε, π.χ. η μετατόπιση των κερδών και βεβαίως υπάρχουν και ανισορροπίες μεταξύ των φορολογικών συστημάτων των κρατών μελών. Αυτά είναι επιβλαβείς πρακτικές και εδώ πέρα νομίζω πρέπει να επιβληθεί σωστά ένας κώδικας συμπεριφοράς και να ενισχύσουμε την σωστή και αποτελεσματική εφαρμογή του κώδικα αυτού συμπεριφοράς. Θέλετε να επανέλθετε. Ε, κύριε Επίτροπε, αναφερθήκατε και στους φορολογικούς παραδείσους και πολλοί συνάδελφοί μας. Ήθελα συγκεκριμένα να σας ρωτήσω εάν θεωρείτε σκόπιμο ε, τον νομοθετικό περιορισμό ή τον αποκλεισμό των υπεράκτιων εταιριών και ε, ε, που έχουν έδρα σε φορολογικούς παραδείσους από το να συμμετέχουν σε διαγωνισμούς δημόσιων συμβάσεων στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι μια πρόταση που έχει ακουστεί από το, ε, και έχει μελετηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ευχαριστώ πολύ. η απάντησή σας ανέφερα ήδη πως ε, θεωρώ πως ε, το ζήτημα της ε, καλής διακυβέρνησης είναι κρίσιμης σημασίας. Θυμάμαι πως όταν ήμουν για πρώτη φορά Υπουργός Οικονομικών στη Λιθουανία, η Λιθουανία δεν ήταν τότε μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οπότε μπορούσα πιο ελεύθερα να παρουσιάσω προτάσεις που είχαν σχέση με τις δραστηριότητες εθνικών εταιριών και υπεράκτιες εταιρείε και εάν θυμάμαι καλά πριν από 10 χρόνια είχαμε επιβάλει την φορολογία στην πηγή για όσους ε, είχαν ε, συναλλαγές με τις λεγόμενες ε, υπεράκτιες εταιρείε. Οπότε νομίζω πώς ε, πρέπει να δούμε το, το ζήτημα αυτό. Δεν είναι εύκολο βεβαίως, αλλά υπό τις συνθήκες της ε, τωρινές, όταν υπάρχει μια παγκόσμια αντίληψη της ε, ζημιάς που προκαλούν η φορολογική παράδοση στα φορολογικά συστήματα των ε, κρατών μελών, ε, των Ηνωμένων Πολιτειών ε, και άλλων χωρών πρέπει να καταλήξουμε σε κάποια κοινή λύση. Ωραία. Ήταν σύντομη ερώτηση, οπότε ήταν κάπως πιο μεγάλη απάντηση. Περνάμε τώρα στον κύριο Ντομενίτση, εκ μέρους των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών. Mr. Senator, λέει Θεωρείτε ότι θα ήταν ρεαλιστικό να προτείνετε μία συζήτηση για ένα κοινό φορολογικό πλαίσιο μεταξύ ε, κρατών μελών πέρα από την εναρμόνιση και την good governance που μας υπενθυμίσατε στην παρέμβασή σας. Απαντώντας το πέμπτο ερώτημα στο ερωτηματολόγιο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, εσείς αναφέρεστε στη δυνατότητα εισαγωγής ενός φόρου για τις χρηματοοικονομικές συναλλαγές. Πότε θα υποβληθεί αυτή η πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και ποιος θα είναι ο συσχετισμός της με άλλες χώρες, διότι και ο πρόεδρος Ομπάμα σκέφτεται κάτι τέτοιο. Ποιος θα είναι ο τελικός σκοπός λοιπόν αυτής ε, της φορολόγησης, δηλαδή εσείς μιλάτε μόνο για χρηματοπιστωτικές συναλλαγές ή επεκτείνεστε και αλλού. Απάντηση επί δύο λεπτά. Αυτό το ζήτημα εξετάστηκε σε πολλά φόρα και υπάρχει η απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου να αποτανθεί στο Διεθνές Νομισματικό Ταμείο για μία ανάλυση ως προς τις ε, πιθανές εφαρμογές αυτού του φόρου σε παγκόσμιο επίπεδο. Αυτή είναι η θέση της Επιτροπής δηλαδή, ότι μπορούμε να κινηθούμε να προωθήσουμε αυτή τη συγκεκριμένη πρόταση εάν εφαρμοστεί παγκοσμίω. Προσωπικά πιστεύω ότι θα πρέπει να προβάλλουμε μία ενδελεχή μελέτη αντικτύπου για ενδεχόμενες επιπτώσεις ως προς τη φορολόγηση των χρηματοπιστωτικών συναλλαγών, διότι υπάρχουν πολλά ερωτηματικά στα οποία δεν έχει δοθεί απάντηση. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε πώς χρησιμοποιούνται τα έσοδα, ποια θα ήταν η βάση αυτής της φορολόγησης και ποιες επιπτώσεις θα έχει στον όγκο συναλλαγών, διότι στις χρηματοπιστωτικές ε, αγορές υπάρχει και μία μελέτη από πλευράς Αυστρίας, αλλά θα πρέπει να επιτελεστεί μεγαλύτερη πρόοδος για να φτάσουμε σε τελική απάντηση, καθώς και ενδελεχής ε, μελέτη αντικτύπου και οι υπηρεσίες της Επιτροπής είναι έτοιμες να αναλάβουν κάτι τέτοιο σε σχέση με την κοινή παγιοποιημένη, μάλλον ενοποιημένη βάση, εσείς θα χρησιμοποιήσετε τις εργασίες αυτές έτσι ώστε να φέρετε σε πέρας αυτό τον φόρο και θεωρείτε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε μία διαβαθμισμένη εφαρμογή με βάση την ενισχυμένη συνεργασία ως προσωμαδοποίηση ορισμένων χωρών σε σχέση με την ενιαία βάση φορολόγησης, διότι στο πέμπτο ερώτημα μιλάτε για καινοτόμους προτάσεις φορολόγησης. Τι εννοείται, ένα λεπτό για την απάντηση. Σε σχέση με το CCCTB, την ε, ενία φορολογική βάση για τις εταιρείες, και τις επιχειρήσεις, νομίζω ότι θα πρέπει να συνεχίσω τις ε, εργασίες του παρελθόντος, έτσι ώστε το CCCTB να είναι ευεργετικό για τις επιχειρήσεις των κρατών μελών και ιδιαίτερα για τις ΜΜΕ των κρατών μελών. Και ζήτησα από τις υπηρεσίες να λάβουν υπόψη ιδιαίτερα τις ΜΜΕ στον τομέα της ενίας φορολογικής βάσης για τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει να προωθήσουμε αυτή την πρόταση το ταχύτερο δυνατόν. σε σχέση με την εφαρμογή σε ορισμένα κράτη-μέλη. Η πρόταση η ίδια θα είναι ε, εθελοντική, προαιρετική. Άρα οι επιχειρήσεις μπορούν να αποφασίσουν επί του CCCTB και να δεχτούν τις ε, προαπαιτήσεις αυτές. Δεν μπορείτε να έχετε πλήρη απάντηση με τρεις ε, συμπληρωματικές. Ε, ο κύριος Σμιτ. Ευχαριστώ κύριε Σιμέτα. Φιλελεύθερος, κάθομαι στο, κέντρο ως φιλελεύθερος. Βρισκόμαστε σε λεπτή φάση της ακρόασης. Φόροι, φόροι. Αυτό ενδιαφέρει όλους τους πολίτες. Είναι ένα αρκοπέδιο για έναν επίτροπο ο ο πρώην Επίτροπος Μόντι, όπως ξέρετε, ετοιμάζει μια έκθεση με συστάσεις για να ξανά ξεκινήσει η ενιαία αγορά και ο καθηγητής Μόντι τονίζει την ανάγκη ενσωμάτωσης στην αγορά μετριάζοντας, περιορίζοντας τον φορολογικό ανταγωνισμό. Περιορισμός του φορολογικού ανταγωνισμού. Ποια είναι η απόψή σας για αυτή τη θέση του κύριου Μόντι και τι πιστεύετε ότι θα βγει από την έκθεση Μόντι και τι ελπίζετε να βγει από την έκθεση αυτή του κυρίου Μόντι. Απάντηση δύο λεπτών. Έχουμε κοινέ αξίες με τον κύριο Μόντι. Όσον αφορά την αγορά. Η πιο μεγάλη επίτευξη της Ένωσης είναι η ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Αλλά δεν είναι τέλεια. Ο στόχος μας και του Επιτρόπου Μπαρνιέ, του υποψήφου Επιτρόπου Μπαρνιέ και άλλων Επιτρόπων και του υποφαινόμενου είναι να κλείσουμε τα παραθυράκια που υπάρχουν σχετικά με την εσωτερική αγορά και σε θέματα φορολογίας έχουμε ακόμα πολλά παραθυράκια. Και ζώντας την κρίση, καλό θα είναι να αντιμετωπίσουμε τα θέματα αυτά. Και όταν μιλάμε για ανταγωνισμό, εγώ θα προτιμούσα συνεργασία των κρατών στα φορολογικά. Αλλά είμαι υπέρ και του θεμητού ανταγωνισμού αρκεί να μην οδηγεί σε καθοδική κίνηση. Γι' αυτό η Επιτροπή πρέπει να παρακολουθεί την κατάσταση, να έχουμε ένα καλό ισορροπημένο επίπεδο φορολογικού ανταγωνισμού, που να είναι εποφελής και για την ανάπτυξη των κρατών μελών διότι αν δεν έχουμε ανταγωνισμό και σε φορολογικά καθόλου, τότε μερικές χώρες μπορεί να προσπαθήσουν να λύσουν όλα τους τα προβλήματα με, μέσω εργαλείων φορολογίας, που δεν είναι θεμητό. Δευτε, δευτερολογία. Φυσικά, αλλά ο θεμητός ανταγωνισμός επιδέχεται πολλές ερμηνείες κατά χώρα. Έχω άλλη μια ερώτηση. Ο κύριος Μόντι δεν αναφέρεται στο επίπεδο της φορολογίας, ενώ οι πολίτες ενδιαφέρονται για το επίπεδο της φορολογίας. Θεωρείτε το επίπεδο γενικά θα πέσει στην Ευρώπη ή θα αυξηθεί λαμβάνοντα υπόψη και τα συνταξιδετικά συστήματα, το δημογραφικό, το πρόβλημα της αυτοκίνητο βιομηχανία, κρατικές ενισχύσεις κλπ. Μπορείτε να κάνετε κάποια πρόβλεψη. Και μια τελευταία ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Οι υπουργοί είναι πολύ στενοκέφαλοι σε αυτό. Δεν πείθονται. Είναι πείσμονες. Πώς θα πείσετε αυτούς τους πείσμενος και ξεροκέφαλος υπουργού οικονομικών. Απάντηση. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος, παρότι η ερώτηση είναι δύσκολη. Το γενικό επίπεδο φορολόγησης στην Ένωση είναι ψηλότερο από ό,τι στις Ηνωμένες Πολιτείες ή την Ιαπωνία, γύρω στο 12% περίπου. Είμαστε μια ένωση με ψηλή φορολογία σχετικά. Από την άλλη μεριά υπάρχουν και άλλα θέματα που τα αναφέρατε. Η κρίση, το πρόβλημα του ανερχόμενου χρέους και η φορολογία είναι ένας χώρος όπου οι κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν διάφορα εργαλεία. Βέβαια, ο πιο καλός τρόπος αντιμετώπιση αυτών των θεμάτων είναι το σκέλος των δαπανών. Και αν χρειαστεί και στο σκέλος των εσόδων. σας ευχαριστούμε. Επόμενος ομιλητής, Ελκ Astrid Λουλίν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, η ερώτησή μου αφορά τους ειδικού φόρους κατανάλωσης, ιδιαίτερα για τα αλκοολούχα ποτά. Στο παρελθόν ο προκάτοχός σας, η Επιτροπή κατ' επανάληψη έσπασε τα μούτρα της, ευτυχώς, σε σχέση με μια πρόταση αύξησης των ειδικών φόρων κατανάλωσης και κατάργηση του συντελεστού 0 για τα για κρασιά. Δεν τρανκίλ. Εσείς σκοπεύετε να προωθήσετε τέτοιου είδους προτάσεις. Ο συντελεστής 0 για το κρασί θα πρέπει να καταργηθεί. Η αύξηση του ελάχιστου συντελεστή από το 92 και μετά δεν οδήγησε σε εναρμόνιση δεν θεωρείτε ότι θα έπρεπε να εισαχθούν και μέγιστοι συντελεστές αντί να αυξάνουμε ή να θέλουμε να αυξάνουμε συνεχώς τον ελάχιστο συντελεστή που και αυτό εμπεριέχει έναν κίνδυνο έντασης του πληθωρισμού. Ευχαριστώ. Απάντηση δύο λεπτών. για τους ειδικού φόρους κατανάλωσης είναι ένας πολύ ενδιαφέρον χώρος και ως πρώην ε, υπουργό Οικονομικών το γνωρίζω το χώρο αυτό. Έχω πάρει πάρα πολλές σχετικές αποφάσεις στη Λιθουανία. Συμφωνώ με τη θέση σας ότι η φύση των ειδικών φόρων κατανάλωσης ε, μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του πληθωρισμού. Και γίνονται συνεχείς προσπάθειες προσαρμογής των ελάχιστων συντελεστών ως προς τον πληθωρισμό. Αλλά εδώ έχουμε και διαφορές στους ειδικούς αυτούς φόρους από χώρα σε χώρα. Ιδιαίτερε χώρε που βρίσκονται στο εξωτερικό σύνορο τη Ένωση και τι γειτονικέ του χώρε. Και η διαφορά, του συντελεστή δημιουργεί ε, όθηση στο λαθρεμπόριο. Πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Γενικά θεωρώ ότι οι εξαιρεσει σε θέματα φορολογίας δεν είναι η καλύτερη λύση. Και αυτό αφορά και κρασί. Βέβαια ξέρω ότι είναι δύσκολο να καταλήξουμε σε μια κοινή αποδεκτή λύση γιατί απαιτείται ομοφωνία. Ελπίζω να ε, σημειωθεί όμως πρόοδος και στο θέμα αυτό εκ μέρους μας. τη δευτερολογία. Κύριε Πρόεδρε, θα συνεχίσει στα γερμανικά. συνεχίσει στα γερμανικά. Νομίζω πως πρέπει να κάνουν πάρα πολλά πράγματα, να ενημερωθούν για πάρα πολλά πράγματα οι επίτροποι, γιατί αυτά τα οποία μας λέτε εδώ πέρα δεν βγάζουν νόημα. Οπότε εγώ θα μπορούσα ευχαρίστως να σας βοηθήσω για να καλύψετε αυτό το έλλειμμα που έχετε στην ε, ενημέρωσή σας. Αλλά δε, δεν μπορείτε να απαντάτε έτσι. Και οπωσδήποτε δεν αντιλαμβάνεστε περί πρόκειται. Έχουμε κοινή αγορά, κύριε Επίτροπε. Δεν έχετε ακούσει ποτέ για φορολογικό ανταγωνισμό τίποτα. One to defend yourself in Ένα λεπτό για να υπερασπιστείτε τον εαυτό σας. Λυπούμε αν ε, η απάντησή μου δεν ε, ήταν ικανοποιητική. Αλλά ανέφερα σε πολλές ε, απαντήσεις πως Είμαι υπέρ ε, της ε, ανάπτυξης ε, της κοινή αγοράς και η φορολογική πολιτική είναι μια πολιτική που θα πρέπει να βοηθήσει στην ανάπτυξη της εσωτερικής αγοράς. Και σκοπεύω να εφαρμόσω τα όσα προτείνονται στις γραπτές μου απαντήσεις. Και τα όσα είπα κατά τη διάρκεια της ακρόασης. Σας ευχαριστώ. Περνάμε στους σοσιαλιστές και δημοκράτες, την κυρία Άλβαρες. Ε, ευχαριστώ κύριε Σεμέτα. Χάρηκα ιδιαίτερα που άκουσα την αδιάσυστη θέση σας ε, για την κατάργηση των φορολογικών παραδείσων και την κατάργηση, την καταπολέμηση της φορολογικής απάτης. Θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την απάτη και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη την αντίσταση ορισμένων κρατών να κινηθούν προς αυτή την κατεύθυνση. Κύριε Σεμέτα, θα ήθελα να καταβληθεί μία προσπάθεια σε σχέση με την οδηγία που προέβαλε ο κύριος Κόβατς για τον φορολογικό συντονισμό. Τι πιστεύετε για την άρση του τραπεζικού απορρίτου και την αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών σαν γενικό κανόνα που να διέπει της χώρας και ποια μέτρα θα προτείνετε έτσι ώστε να τηρηθεί αυτή η οδηγία ή για την μη τήρηση αυτής της οδηγίας, την ενδεχόμενη μη τήρησή της. Έχετε δύο λεπτά για να απαντήσετε. Ναι. Νομίζω πως είναι πολύ σημαντικό να περάσει η νομοθεσία στον τομέα της ε, φορολογικής ε, συνεργασίας. Και εδώ νομίζω πως το ζήτημα της αυτόματης ανταλλαγής ε, πληροφοριών είναι κρίσιμο. Και δεν έχω αμφιβολία, τους πρέπει να προχωρήσει. Θα ξέρετε πως ε, σημειώσαμε πρόοδο στην διαπραγμάτευση αυτής της πρότασης και υπάρχουν δύο κράτη-μέλη ακόμα τα οποία εξακολουθούν να είναι κατά αυτής της πρότασης και θέλουν μια προσέγγιση πακέτο δηλαδή και συμφωνίες με το Λιχνεστάιν και άλλες μικρές χώρες στην Ευρώπη. Και το θεωρούν αυτό προαπαιτούμενο αλλά νομίζω πως ε, το ΕΚΟΦΗΝ ήδη της 19ης Ιανουαρίου θα συνεχίσει την συζήτηση επ' αυτού του ζητήματος. Και ελπίζω πως ε, τα δύο αυτά κράτη-μέλη θα πιστούν να μην μπλοκάρουν την απόφαση αυτή γιατί νομίζω πως είναι και για αυτές τις χώρες σημαντικό ε, να υπάρχει αυτόματη ανταλλαγή πληροφοριών. Δευτερολογία, κύριε Άλβαρης. Ευχαριστώ, κύριε Σεμέτα. Και εμείς θα σας υποστηρίξουμε για να προχωρήσετε προς αυτή την κατεύθυνση. Όπως είπατε, είναι η κατάλληλη στιγμή για να γίνει κάτι τέτοιο και ο Ευρωπαίος πολίτης δεν κατανοεί όταν δεν υπάρχει αυτή η αυτόματη ανταλλογή έτσι ώστε να εναρμονίσουμε τα ε, φορολογικά συστήματα και την άρση του απορρίτου. Γι' αυτό σας ευχαριστώ για την απάντηση. Ε, ε, δεν νομίζω ότι πρέπει να απαντήσετε εκτός αν το θέλετε διακαώς. Όχι, εντάξει. Σε αυτή την περίπτωση ε, εξ μάλλον ο κύριος Φέρμπερ έχει το λόγο εξ του ΕΛΚ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κύριε υποψήφιοι επίτροπε. Ακούσαμε πάρα πολλά πράγματα για την καταπολέμηση της απάτης ε, και τη φορολογία, αλλά δεν είστε μόνο γι' αυτό υπεύθυνος, γι αυτό υπεύθυνος αλλά και για το φορολογικό δίκαιο. Και έχουμε κάποια ζητήματα που χρήζουν εναρμόνισης, ε, υπεραιτέρω εναρμόνιση. Θα αναφέρω κάποια πραγματάκια πρώτα απ' όλα η ο τόπο επιμέτρησης φορολογικής βάσης ε, στη φορολογία των επιχειρήσεων και βέβαια υπάρχει και το ζήτημα της μεταρρύθμισης του ΦΠΑ. Συγκεκριμένα λοιπόν θα ήθελα να ακούσω πότε σκοπεύετε να καταθέσετε προτάσεις, γιατί χωρίς προτάσεις τη Κομισιόν και με τη Λισαβόνα δεν ε, γίνεται τίποτα. Ευχαριστώ. Η απάντησή σας. Για την ε, κοινή ενοποιημένη φορολογική βάση. Η Κομισιόν θα καταθέσει πρόταση το συντομότερο δυνατόν. Πρέπει να τελειώσει η αξιολόγηση αντικτύπου κάποιων στοιχείων και όταν ολοκληρωθεί αυτή αυτή η αξιολόγηση ε, ελπίζουμε πως θα κατατεθεί και η πρόταση αυτή. Εγώ σκοπεύω οπωσδήποτε να το ξεκινήσω, αλλά είναι απόφαση του σώματος των επιτρόπων. Οπότε πρέπει να αποφασίσει συνολικά η Επιτροπή. Εάν κατάλαβα καλά, επίσης με ρωτήσατε για τη μεταρρύθμιση του ΦΠΑ. Η πρόθεσή μου είναι να αναπτυχθεί μια νέα στρατηγική ΦΠΑ που θα αντιμετωπίσει τα ζητήματα που ευσεκρεμεί η προηγούμενη στρατηγική και θα ασχοληθεί και με τα ζητήματα ενός οριστικού συστήματος ΦΠΑ και της μελλοντικής ανάπτυξης ενός τέτοιου συστήματος που θα λαμβάνει υπόψη την προηγούμενη στρατηγική και το ότι πλέον χρειαζόμαστε ένα νέο όραμα. Στην αρχή νομίζω λοιπόν της ιτίας μας θα καταθέσουμε προτάσεις για τη νέα στρατηγική του ΦΠΑ δευτερολογία. Ναι, ευχαριστώ. Να παραμείνω στον ΦΠΑ. Ο Επίτροπος Μόντι είχε πει όταν, ιδρύθηκε, όταν συστάθηκε η εσωτερική αγορά πως το 1996 θα έπρεπε να ισχύει μέχρι το 1996 πλέον η αρχή Τη χώρα προέλευση των ΦΠΑ. Το 96 έχει παρέλθει, ο κύριο Μόντι δεν είναι πια εδώ πέρα. Πότε σκοπεύετε να μπορέσετε να εφαρμόσετε κάτι τέτοιο. Ε, ένα λεπτό για την απάντηση. Γνωρίζετε πως ε, αυτή τη στιγμή έχουμε μεταβατικά συστήματα ΦΠΑ και το σύστημα είναι σε μεταβατική φάση εδώ και πολύ καιρό. Η νέες αποφάσεις ε, στον τομέα της φορολογίας ειδικά όσον αφορά τον ΦΠΑ των υπηρεσιών πηγαίνουν ε, προς την ε, αρχή μάλλον του προορισμού παρά της προέλευσης. Και στην στρατηγική των νέων εξελίξεων στον τομέα του ΦΠΑ σκοπεύω να ασχοληθώ με αυτό το ζήτημα. Σας ευχαριστώ. Τελειώνουμε έτσι με το κομμάτι της Επιτροπής Οικονομικών Ζητημάτων και θα δώσω τώρα την Προεδρία στον Μάλκομ Χάρμπορ για να περάσουμε στην Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κυρία Μπόλς και ευχαριστώ που μας δίνετε την ευκαιρία. Για να προσδιορίσουμε την ακρόαση θα ήθελα να πω ότι από πλευράς εσωτερικής αγοράς μας ε, ενδιαφέρει η πολιτική σας κύριε Επίτροπε ως προς την Τελωνιακή Ένωση. Με βάση τη θητεία σας βλέπουμε ότι ε, ότι η Τελωνιακή Ένωση αφορά την καλύτερη διαχείριση, βέλτιστη διαχείριση και καλύτερο συντονισμό σε αυτό το τομέα. Ε, χαίρομαι διότι παρευρίσκονται πολλά μέλη της ε, Επιτροπής μας για να σας υποβάλουν ερωτήσεις. Ο πρώτος ομιλητής, η πρώτη ομιλήτρια μάλλον είναι η κυρία Κορχόλα και μετά Στάιλερ και θα ακολουθήσουμε ακριβώς την ίδια αρχή, δηλαδή ένα λεπτό, δύο λεπτά, ένα και ένα λεπτό αντιστοίχως. Κοχόλα. Οι περισσότεροι από εμά κατανοούν ότι θα πρέπει να μειωθούν οι εκπομπές μέσα στα πλαίσια της πράσινης φορολόγησης και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια κοινή προσέγγιση. Πιστεύω λοιπόν ότι δεν θα πρέπει να πληγούν ε, τα κράτη τα οποία δεν προβαίνουν σε dumping εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει και το πρόβλημα του θέμη του ανταγωνισμού και η κατάσταση μπορεί να επιδεινωθεί αν η Συμφωνία της Κοπενχάγης σημαίνει ότι θα πρέπει να ορίσουμε το στόχο μας όχι το 2020 αλλά το 2030. Μιλήσαμε για τη φορολόγηση του άνθρακα πολλές φορές. Η Επιτροπή θα προτείνει έναν κοινό φόρο. Θεωρείτε ότι η κοινή φορολόγηση θα ήταν ευεργετική λαμβάνοντας υπόψη και τις εμπορικές μας σχέσεις καθώς και τη θέση μας στην παγκόσμια αγορά. Πιστεύετε ότι θα πρέπει να ορίσουμε τον στόχο όχι στο 2020, στο 2030 και θεωρείτε ότι υπάρχουν, έχουν γίνει αρκετές έρευνες και ποιες θα μπορούσαν να ήταν οι συνέπειες. Πριν ε, απαντήσει ο κ. Σεμέτα θα ήθελα να επικρατήσει ησυχία στην αίθουσα και θα ήθελα να σας, ε, μιλήσω, να σας ε, υπενθυμίσω ότι μιλάμε για την Τελωνιακή Ένωση. Θα μπορούσατε να περιορίσετε τις ε, ερωτήσεις σας στο τομέα που μας αφορά. Η κυρία Κοχόλα δεν μπορεί να υποβάλει συμπληρωματική γιατί επεκτάθηκε πολύ. Σε μέτα. Ευχαριστώ πολύ για την ερώτησή σας. Βρισκόμαστε στο τομέα της φορολόγησης και νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλη σημασία να δούμε πώς θα προωθήσουμε την πράσινη φορολόγηση, πώς να την ενισχύσουμε με βάση την οδηγία για την φορολόγηση της ενέργειας. Αυτή η οδηγία θα είναι από τις πρώτες μου προτεραιότητες στη μελλοντική μου εργασία υπό τον όρο ότι θα εγκρίνεται την εντολή και τη θητεία μου. Και βεβαίως αυτή η οδηγία για τη φορολόγηση της ενέργειας συμπεριλαμβάνει και την φορολόγηση του διοξιδίου του άνθρακα, διαχωρίζει δηλαδή την ενεργειακή φορολόγηση ως προς το σκέλος της ενέργειας και το σκέλος του διοξιδίου του άνθρακα. Κάτι το οποίο θα μας βοηθήσει να ορίσουμε μια σωστή φορολόγηση ως προς τον τομέα του άνθρακα, ο οποίος δεν καλύπτεται από το σύστημα ε, ανταλλαγής και φορολόγησης εκπομπών. Ως προς τη διασυνοριακή, τις διασυνοριακές διαρροές, αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό ζήτημα και θα προτιμούσα να ληφθούν υπόψη διεθνείς συμφωνίες οι οποίες θα επιτευχθούν σε αυτό το τομέα, αλλά η Επιτροπή μελετά αυτή τη στιγμή τους αντικτύπους της ε, κατάστασης και όταν ε, διεκπαιρεωθεί αυτή η μελέτη θα υποβάλω προτάσεις σε αυτό το τομέα αν κάτι τέτοιο κρυθεί αναγκαία. Ευχαριστούμε πολύ, ε, Στάιλερ. Όχι, όχι, κυρία Κορόλα δεν ε, μπορεί να δευτερολογήσει, γιατί δεν υπέβαλε ερωτήσει ω προ την Τελωνιακή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σεμέτ. Σε σχέση με το σχέδιο μη παραχαράξεων, καταπολέμηση των παραχαράξεων, υπάρχει παραχάρηξη ε, φαρμακευτικών σκευασμάτων τα οποία θα μπορούσαν να ε, οδηγήσουν και στο θάνατο πολιτών. Επειδή μιλάτε για την παραχάρεξη ε, φαρμακευτικών παρασκευασμάτων, ε, θεωρείτε ότι θα πρέπει να ενταχθεί, μπορείτε μάλλον να μου εγγυηθείτε ότι κάτι τέτοιο θα ενταχθεί στο σχέδιο δράσης καταπολέμησης παραχάραξης. Σε μέτα. Ευχαριστώ το θέμα της ε, παραχάραξης είναι ύψης της σημασίας στα πλαίσια του χαρτοφυλακίου μου και θα εφαρμόσω τάχιστα το πρόγραμμα δράσης 2009-2012 κατά της ε, παραχάραξης όπου εντάσσονται διατάξεις ε, σχέση με τροποποίηση της νομοθεσίας ως προς ε, επιχειρησιακά ζητήματα συνεργασίας με τις φαρμακοβιομηχανίες. Θα εξετάσω όλες τις επιμέρους θέσεις έτσι ώστε να επιτελεστεί πρόοδο στο θέμα καταπολέμησης της παραχάραξης και ιδιαίτερα ως προς τα φαρμακευτικά σκευάσματα. Κάτι τέτοιο είναι επώδυνο και επικίνδυνο για τον πολίτη η παραχάραξη αυτή και θα πρέπει να αποτιμήσουμε και τους κινδύνους. διότι πρόκειται για επιζήμια σκευάσματα, επιζήμια για την υγεία του πολίτη. Γι' αυτό θα συνεργαστώ μαζί σας σε αυτό το τομέα. Η δευτερολογία. Ευχαριστώ. Αναφέρατε ότι το πρόγραμμα δράσης ισχύει μέχρι το 2012. Τι θα γίνει μετά το 2012, πώς θα προωθηθεί αυτό το σχέδιο δράσης κατά της παραχάραξης. Νομίζω ότι ένας βασικός τομέας είναι να φτάσουμε σε διεθνείς συμφωνίες ως προς την καταπολέμηση της παραχάραξης. Ήδη έχουν συναυθεί συμφωνίες και μία πολύ πρόσφατα ε, συνήφθη με την Κίνα. Αλλά νομίζω ότι η παραχάραξη είναι παγκόσμιο ζήτημα, δεν αφορά μόνο τον τελωνιακό τομέα. Άρα, για το μέλλον θα πρέπει να αναπτύξουμε ένα κοινό πρόγραμμα δράσης έτσι ώστε να συμμετέχουν και οι διεθνείς φορείς καθώς και ε, άλλα θεσμικά όργανα που σχετίζονται με το θέμα της παραχάραξης έτσι ώστε να έχουμε συντονισμένες προσπάθειες σε παγκόσμιο επίπεδο ως προς τα παραχαραγμένα προϊόντα και αγαθά. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Κάμπ και η κυρία Σαλτεμόζα μετά. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Κύριε Πρόεδρε, έχω ερώτηση για τη σχέση μεταξύ ΟΛΑΦ και της Γενικής Διεύθυνσης Φορολογίας και Τελωνιακής Ένωσης. Μιλήσαμε για τον πρόεδρο του Όλαφ, αλλά η ομάδα μου, το ΕΛΚ, θεωρεί πως υπάρχουν κάποια προβλήματα στο χαρτοφυλακείο σας για τις αρμοδιότητες του Όλαφ αφενός και της Γενικής Διεύθυνσης Τελωνίων απ' την άλλη. Πώς θα διαχειριστείτε αυτές τις δύο αρμοδιότητες ε, στην πράξη. Αυτό είναι το ερώτημά μου κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε. Ευχαριστώ. Από ό,τι κατάλαβα μιλάτε για πιθανά συγκρόμενα συμφέροντα στο αξίωμα μου. Σας διαβεβαιώ πως ε, δεν βλέπω τέτοια πιθανότητα συγκρόμενων συμφερόντων ε, εντό ε, του χαρτοφυλακίου δηλαδή μεταξύ Όλαφ και Γενική Διεύθυνση ε, Φορολογία τη Τελωνιακή Ένωση, γιατί η ευθύνη τη Γενική Διεύθυνση είναι η ανάπτυξη νομοθεσία και η παρακολούθηση της εφαρμογής της νομοθεσίας, ενώ η νομοθεσία κάθε αυτή εφαρμόζεται από τα κράτη-μέλη και είναι και προς το συμφέρον της ε, Γενικής Διεύθυνσης ε, να καταπολεμήσει την ε, απάτη και η καταπολέμηση της απάτης είναι αν θέλετε αυτό το οποίο διέπει όλο μου το, το χαρτοφυλάκιο και συνδέει τα διάφορα τμήματα αυτά που φορούν τη φορολογία, τα τελωνία και τις πάνε το πώς ξοδεύονται τα ευρωπαϊκά κονδύλια. Οπότε δεν νομίζω πω υπάρχει ζήτημα σύγκρουση συμφερόντων συμφεροντων εντο του χαρτοφυλακίου μου. Εάν δούμε την ε, τρέχουσα σύνθεση του χαρτοφυλακίου, εκεί όπου υπάρχει εσωτερικός έλεγχος ε, και η διοίκηση σε ένα χαρτοφυλάκιο, εκεί είναι πολύ πιθανότερος ο κίνδυνος ε, σύγκρουση συμφερόντων από ότι στο δικό μου χαρτοφυλάκιο. Κύριε Φαντεκάμπ, ευχαριστώ. Κύριε Πρόεδρε, με αυτό ακριβώς λέω. Εάν λέει ο κύριος Επίτροπος πως η Ταξούντ καταπολεμά την απάτη και εντωμεταξύ ο Όλαφ, ε, παραδείγματος χάριν, επίσης ασχολείται με αυτό το συγκεκριμένο κομμάτι της απάτης, ποια η σχέση μεταξύ των, ε, των δύο ερευνών και ε, ποια θέση θα, θα πάρετε εσείς. Η απάντηση είναι θα πρέπει να φροντίσουμε να υπάρχει σωστή συνεργασία στην καταπολέμηση της απάτης. Έχουμε συστήματα ανταλλαγής πληροφοριών για θέματα απάτης. Τι μέτρα λαμβάνονται είτε από την Όλαφ είτε από την Ταξούντ και θα πρέπει να γίνει και συντονισμός να μην έχουμε επικάλυψη δύο φορές το ίδιο πράγμα. και μη σωστή χρήση των πόρων. Μέχρι στιγμής στο θέμα αυτό δεν είχαμε προβλήματα και πιστεύω ότι η κατάσταση θα συλλογιστεί θετικά έτσι. Ε, κυρία Μόζα η κυρία Σάλντερ Μόζα ως μέλος της Επιτροπής Εσωτερικής Αγοράς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Επίτροπε, μας είπατε στη γραπτή σας απάντηση ότι για την τελωνιακή πολιτική προέχει η ασφάλεια του καταναλωτή. Και στην απάντηση στην κυρία Στάιλερ είπατε ότι πρέπει να γίνει η καταπολέμηση των απομιμήσεων. Τι θα κάνετε συγκεκριμένα για να έχουμε καλύτερο διάλογο με την Κίνα, την Ιαπωνία, τις Ηνωμένε πολιτειε ιδιαίτερα όσον αφορά την ασφάλεια του πολίτη έναντι των απομιμήσεων. Απάντηση. Είχαμε σημαντική πρόοδο στις σχέσεις Ένωση-Κίνα. Ίσως λίγο λιγότερο με τη Ρωσία. Πιστεύω ότι υπάρχει δυνατότητα να διαπραγματευτούμε και να καταλήξουμε σε συμφωνία με τη Ρωσία Για uh, uh, τις πρόδρομες ουσίες φαρμάκων κλπ. Για την Κίνα υπάρχει συμφωνία συνεργασίας και έχουμε πολύ καλά προγράμματα για πιο, ε, πιο έξυπνους τρόπους μεταφοράς, έγκριση οικονομικών οργανισμών προς αμοιβαία αναγνώριση. προκειμένου να ενισχυθεί το σκέλος της προσφοράς και να έχουμε ασφαλή ανεφοδιασμό όσον αφορά την προσφορά πάντα. Αυτό είναι ένα, ένα ένας τομέας κλειδί για την Επιτροπή. Επερώτηση. Και εγώ θεωρώ ότι και πολλά έχουν γίνει, αλλά τα επικίνδυνα εμπορεύματα που έρχονται στην Ένωση είναι όλο και πιο πολλά. Τι θα κάνετε με τους άλλους επιτρόπους σχετικά με το πρόβλημα αυτό. Τα προϊόντα που έρχονται στην ευρωπαϊκή αγορά δηλαδή να είναι ασφαλή. Πώς θα συνεργαστείτε με τους άλλους επιτρόπους. Απάντηση. Έχετε δίκιο. Το θέμα αυτό αφορά παραπάνω από έναν επιτρόπους. Και πολλές γενικές διευθύνσεις. Θα δούμε με τους νέους επιτρόπους πώς θα αντιμετωπιστεί το θέμα αυτό. Φερρυπίν θα μπορούσαμε να έχουμε μια ομάδα ή ομάδες ad hoc για συγκεκριμένα θέματα, ομάδες επιτρόπων εννοώ. για τις ε, απομιμήσεις ε, το θέμα των πνευματικών δικαιωμάτων, δικαιωμάτων ιδιοκτησίας. θα μπορούσαμε να έχουμε μια ομάδα η οποία να συντονίζει τις δραστηριότητες προτείνοντας συγκεκριμένα μέτρα και πολιτικές. Πρόεδρος, η κυρία Μπαστός, ΕΛΚ. Ευχαριστώ θα επανέλθω στο θέμα της παραχάραξης που μου φαίνεται πολύ σημαντικό που πλήττει την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη της αγοράς και ιδιαίτερα ως προς τα φαρμακευτικά σκευάσματα ε, θέτει σε κίνδυνο τη ζωή των πολιτών και έχει αρνητικές επιπτώσεις στην ευρωπαϊκή οικονομία. Σχετίζεται άμεσα και με το τελωνιακό καθεστώς προβλέπει η Επιτροπή νέες πρωτοβουλίες ε, για την καταπολέμηση της παραχάραξη, παραχάραξης, διότι τα μέτρα που αναφέρεται είναι ε, ευρεία εμβέλειας, δεν είναι συγκεκριμένα. Θα ήθελα να είσαστε πιο συγκεκριμένος ως προς τα μέτρα που θα εισαγάγετε και ποιο θα είναι το χρονοδιάγραμμα εισαγωγής αυτών των μέτρων ως προς τον τελωνιακό κώδικα τι συνοδευτικά μέτρα θα λάβετε ως προς το φορολογικό καθεστώς. Τέλος, ε, προβλέπετε προβλήματα σε σχέση με την εκτέλεση του κανονισμού. Ευχαριστώ. Ε, απάντηση. Ευχαριστώ πολύ. Είπα απαντώντας σε προηγούμενες ερωτήσεις ότι τα θέματα, των, το πρόβλημα των απομιμήσεων και των πλαστών προϊόντων δεν ευθύνει μόνο ενός επιτρόπου αυτού που είναι υπεύθυνο για τα τελωνία. Είναι πολύ ευρύτερο θέμα και χρειάζεται συνεργασία μεταξύ των επιτρόπων. Όσον αφορά το τελωνιακό σκέλος, όταν, κάνουμε, ε, όταν εισάγουμε συστήματα ανάλυσης του κινδύνου θα πρέπει να προσέξουμε ιδιαίτερα το θέμα αυτό των, ε, των απομιμήσεων. και να έχουμε καλύτερη ροή πληροφοριών μεταξύ των εθνικών αρχών. σχετικά με το λαθρεμπόριο τέτοιου είδους ε, προϊόντων. Υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Τώρα για τους τελωνιακούς κώδικες και την εφαρμογή τους. Πραγματικά αυτό είναι μια μεγάλη πρόκληση. Αλλά είναι προς το κοινό μας συμφέρον να εφαρμοστούν μέχρι το 2013 γιατί υπάρχουν πολλοί όροι στους ε, τελωνιακούς κώδικες που μας επιτρέπουν να απλοποιήσουμε τη διαδικασία για τις επιχειρήσεις το χρήση ηλεκτρονικών μεθόδων στα τελωνιακά ή επίσης η διαδικασία του ενιαίου παράθυρου που τη λέμε single window. Η κυρία Μπαστός δευτερολογία. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να μου πείτε το εξής. Ε, είπατε ότι υπάρχουν και άλλοι επίτροποι που είναι υπεύθυνοι στον τομέα της χάραξης. Κατά πόσο θα συνεργαστείτε για να επιτευχθεί μια, ένα συντονισμός για την καταπολέμηση της παραχάραξης και των απομιμήσεων. Είχαμε πολλές ε, συναντήσεις και σεμινάρια στα πλαίσια της ε, νέας Επιτροπής πριν από τις ακροάσεις όπου συζητήσαμε θέματα συντονισμού, μελλοντικού συντονισμού των μελλοντικών δραστηριοτήτων και συμφωνήσαμε, όπως σας προείπα, να προβούμε στη σύσταση ομάδων ad hoc για ειδικά ζητήματα και νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. δηλαδή η συνεργασία στον τομέα της εσωτερικής αγοράς, ε, τελωνιακών ζητημάτων και φορολογικών και άλλων επιτρόπων που θα μπορούσαν να συντονίσουν αυτή τη δράση. Ο κύριος Κρόιτσμαν, που είναι ο τελευταίος ε, ομιλητής ε, από την εσωτερική αγορά. Κύριε Υποψήφιε Επίτροπε, συζητήσαμε για προϊόντα πλαστογραφημένα που μπαίνουν στην ευρωπαϊκή αγορά και γνωρίζετε πως υπάρχουν και εισαγόμενα αγαθά στην ευρωπαϊκή αγορά που δεν εκπληρώνουν τις προδιαγραφές ασφαλείας τι σκοπεύετε να κάνετε για να συντονιστούν τα ευρωπαϊκά τελωνία καλύτερα για την υποκτία της αγοράς για να μην μπαίνουν επικίνδυνα προϊόντα στην αγορά. Δεν θεωρείτε επίσης πως ε, πρέπει να υπάρχει μια ευρωπαϊκή εποπτεία της ε, αγοράς και μια κατανομή των βαρών μεταξύ των κρατών μελών καθώς κάποια κράτη-μέλη φύστανται υπερβολικά μεγάλος, ε, μεγάλο βάρος. Π.χ. να δώσω ένα παράδειγμα, όταν έρχονται στα λιμάνια, π.χ. στο Αμβούργο ή οπουδήποτε αλλού, είναι πάρα πολύ μεγάλος ο φόρτος των ε, τελωνιακών αρχών που πρέπει να διασφαλίσουν την υποπτία της αγοράς και από εκεί πέρα μπαίνουν σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση τα προϊόντα. Κύριε Επιτροπέ, ναι, ευχαριστώ. Ο τελωνιακός ε, κώδικας είναι σύγχρονος, μας δίνει ε, πάρα πολύ καλή ευκαιρία ε, για να σημειώσουμε σημαντική πρόοδο σε αυτό τον τομέα και να έχουμε ένα κεντρικό σύστημα clearing το οποίο αυτή τη στιγμή αναπτύσσεται. Και ε, νομίζω θα επιφέρει επανάσταση στον ε, τομέα αυτόν γιατί όταν εφαρμοστεί ο κάθε έμπορος δεν θα χρειάζεται να μετακινείται με τα αγαθά του που μπαίνουν αυτά στην εσωτερική αγορά αλλά θα υποβάλει τα σχετικά έγγραφα στο οικείο τελωνίο και θα μπορέσουμε να έχουμε και ένα τέτοιο σύστημα και στον τομέα του ΦΠΑ, των δικών φόρων κατανάλωσης, για να έχουμε ένα πραγματικά κεντρικό σύστημα εκαθάρισης ε, συμψηφισμού για όλους αυτούς τους τομείς, έτσι ώστε οι έμποροι να μπορούν ε, να ασχολούνται και να έρχονται σε επαφή με τις αρχές στην πατρίδα τους. Και μάλιστα τα, τα έργα αυτά απαιτούν πάρα πολύ συνεργασία και συντονισμό από τα κράτη-μέλη. Και νομίζω πως ε, με την εφαρμογή αυτή και την παρακολούθηση της ε, προόδου στα έργα αυτά θα διασφαλιστεί ο καλύτερος συντονισμός ε, των θεσμικών οργάνων που εργάζονται και στον τομέα των τελωνιακών, αλλά και σε άλλους τομείς που σχετίζονται με το διεθνές εμπόριο. Κύριε Έχουμε διαφορετικά συστήματα επίβλεψης. Π.χ. στη Γερμανία είναι τα κρατήδια υπεύθυνα για την επίβλεψη. Σε άλλες χώρες είναι κεντρικό το σύστημα. Η επίβλεψη της αγοράς λοιπόν είναι διαφορετική. Υπάρχουν κάποιες αδυναμίες. Τι σκοπεύετε να κάνετε για να υπάρξει βελτίωση στις χώρες όσον αφορά την επιτήρηση της αγοράς. Ναι. Βεβαίως δεν μπορούμε να παρέμβουμε στα εσωτερικά των κρατών μελών. Τα κράτη-μέλη είναι ελεύθερα να φτιάξουν τα συστήματά τους όπως ε, νομίζουν ε, εκείνα. Στόχος μας είναι παρά την ε, ποικιλία των συστημάτων να καταλήξουμε σε κάποιον συντονισμό και νομίζω οι εξελίξεις και η ανάπτυξη της πληροφορικής μηχανογράφησης είναι το μέσο που θα μας επιτρέψει να έχουμε συντονισμό μεταξύ των αρχών των κρατών μελών και να διευκολύνουμε αυτές τις εξελίξεις. Βέβαια υπάρχουν διάφορες σκέψεις για κάποια έτσι, κοινά τελωνία, αλλά αυτό ανήκει στο μέλλον παρά στο παρόν της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ τους συναδέλφους και τον Επίτροπο. Θα ήθελα τώρα να παραδώσω ξανά την Προεδρία στον Πρόεδρο της Επιτροπής Ελέγχου του Προπολογισμού. Ευχαριστώ τον Πρόεδρο Χάρμπερ. Θα δώσω το λόγο στον υποψήφιο Επίτροπο για μια τελευταία σύνοψη θέση, αν θέλει, μερικών λεπτών. So, thank you very Σας ευχαριστώ για τις ερωτήσεις που μου υποβάλατε κατά τη διάρκεια αυτής της ακρόασης και νομίζω ότι αυτό είναι ο πραγματικός, ένας πραγματικός διάλογος μεταξύ των αντίστοιχων κοινοβουλευτικών επιτροπών και εμού. Νομίζω ότι ο ανοιχτός αυτός διάλογος είναι ύψης της σημασίας έτσι ώστε να επιλύσουμε ζητήματα και προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν βρίσκομαι σε πολύ ευχάριστη, ας το πούμε, εύκολη θέση, διότι έχω να συνεργαστώ με τρεις επιτροπές αλλά νομίζω ότι ε, υπήρξε αγαστή συνεργασία με την προηγούμενη Κοινοβουλευτική Επίτροπη, διότι όπως ξέρετε είμαι υπεύθυνο ήμουν υπεύθυνο για θέματα προϋπολογισμού και θα χρησιμοποιήσω την πείρα μου αυτή συνεργασίας και συνεργατικής διάθεσης για την ε, περαιτέρω συνεργασία με την Επιτροπή Ελέγχου Προϋπολογισμού Εσωτερικού, Εσωτερικής Αγοράς και Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων. Σήμερα άκουσα πολύ ενδιαφέρουσες ε, ε, ερωτήσεις που θα με οδηγήσουν σε νέες ιδέες και νέες προτάσεις για το μέλλον και υπάρχουν πολλά ζητήματα τα οποία θα πρέπει να επιληθούν στα θέματα νέων δαπανών. Είμαι έτοιμος να συνεργαστώ μαζί σας. Θα προταθούν ε, νέα πλαίσια και χρειάζομαι τη δική σας πλήρη υποστήριξη κατά τις συζητήσεις κατά την επίτευξη συμφωνιών για να προωθήσουμε αυτές τις προτάσεις. Στο τομέα της φορολόγησης και τον τελωνιακό τομέα η κατάσταση είναι πιο δυσχερής. Στο τομέα της φορολόγησης χρειαζόμαστε ομοφωνία για τη λήψη αποφάσεων και εδώ θα βασιστώ στη δική σας υποστήριξη όταν ανακύψουν νέες προτάσεις που θα αφορούν την εσωτερική αγορά, την καταπολέμηση των φορολογικών παραδείσων και την εφαρμογή της πράσινης φορολόγησης. Νέες προτάσεις λοιπόν και οι ιδέες προβάλλονται, βρίσκονται εν εξελίξη και θα βρίσκομαι σε στενή συνεργασία με σας, δέχομαι κάθε ιδέα, ανταλλαγή απόψεων για ζητήματα που άπτονται του χαρτοφυλακίου μου και νομίζω ότι η συνεργατική αυτή διάθεση θα μας βοηθήσει να λάβουμε τις αποφάσεις που θα βοηθήσουν την αναπτυξιακή πορεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σας ευχαριστώ πολύ.